Buenos días, colegas. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα το πρωί αλλά και ενδιαφέρουσα. Αρχίζουμε με ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές ε, του ΟΙΕ στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Θα μιλήσουμε για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να καλωσορίσω εδώ την κυρία Σουλτανόγλου που είναι αναπληρωτής ε, Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και παρακολουθεί τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών και είναι διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΗΕ. Συνοδεύεται από τους συντονιστές του ΟΗΕ των έξι χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι ο κύριος Χάρς, την Ουκρανία ο κύριος Βόκερ, Μολδαβία η κυρία Αντώνια Ναφίνα Κατσέβα, Γεωργία. Ντονιέλ Σκοτ, Αρμενία, ο κύριος Τεπράλης Μπουσέτο, Αζερβαϊτζάν, ο κύριος Δονοτόνιος Φράκ. Οι συντονιστές είναι πρέσβεις των Ηνωμένων Εθνών επιτόπου, γιατί ζουν στις χώρες αυτές. Και εκεί φροντίζουν για τον συντονισμό των δράσεων των Ηνωμένων Εθνών και για τα προγράμματα των διαφόρων υπηρεσιών. Εκπροσωπούν τον ΟΗΕ σε όλες του τις διαστάσεις και έχουν επαφές εκ μέρους του ΙΕ με όλες τις αρχές εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μα λοιπόν να μάθουμε ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνουν τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτές τις χώρες, ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς βλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη την κατάσταση επιτόπου. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε πρώτα ανατολικά της Ουκρανίας ποια είναι η κατάσταση δεδομένων των πολεμικών φωνών τον τελευταίο καιρό και να δούμε πώς προχωρά το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Επίσης θα θέλαμε να αξιολογήσετε με ειλικρίνεια και αν χρειάζεται να είστε και επικριτικοί στη συμπληρωματικότητα των δράσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΙΕ και να μας πείτε ποιες είναι οι δυναμίες και να μας κάνετε και προτάσεις για να βελτιώσουμε τη δράση μας. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε τις απόψεις σας για το πόσο καλή είναι η πολιτική μας ανατολικής γειτονίας και πόσο βοηθάει τη δράση του ΟΙΕ. Προτείνω η ανταλλαγή απόψεων να λάβει χώρο εξή. Πρώτον, η κυρία Σουλτάνογλου να μας παρουσιάσει τις δράσεις και τις προτερότητες του ΟΙΕ σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας και στη συνέχεια να ακούσουμε τους συντονιστές που ζουν εκεί να συμπληρώσουν την παρουσίαση αυτή και να μας παρουσιάσουν ειδικά στοιχεία που πιστεύουν ότι είναι σημαντικά για τις χώρες όπου ζουν. Μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κυρία Σουλτάνογλου, έχετε το λόγο. Έχετε 5-7 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτήν την όμορφη εισαγωγή και σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε να έρθουμε και να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Χαιρετίζω λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά τους αξιότιμους ευρωβουλευτές και ήρθα εδώ με τους συναδέρφους μου για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Και είναι προνόμιο για μας που σας συναντούμε και που έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΟΗΕ και τις απόψεις του ΟΗΕ όσον αφορά τις αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Ήδη ο πρόεδρος παρουσίασε τους έξι εκπροσώπους, πέντε ουσιαστικά, γιατί ο εκτός δεν ήταν πολύ καλά σήμερα και δεν μπόρεσε να έρθει, είναι εκείνο που βρίσκεται στη Λευκορωσία κανονικά. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την επιθυμία του Πρόεδρου σας για καλή καρποφόρα συζήτηση σήμερα το πρωί για τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και για τις σχέσεις μας στην περιοχή. Ένας από τους λόγους που ήρθαμε εδώ τόσο πολύ είναι επειδή είχαμε πρόσκληση από τον Κρίστιαν Τέλσαν, από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΡ, προκειμένου να συζητήσουμε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική της Ανατολικής Γειτονίας. Θα συναντηθούμε μαζί του σήμερα κάποια στιγμή αργότερα και θα ανταλλάξουμε απόψεις μαζί του για την πολιτική αυτή. Οπότε ήδη μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήθελε να συζητήσει μαζί μας. Τώρα, η προβληματική τομεί όσον αφορά την πολιτική αυτή, οι δικοί σας, έχουν να κάνουν και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως ΟΙΕ εκεί. Την βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση, τη διαφάνεια, την λογοδοσία, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ενέργεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, επικεντρωνόμενη ιδιαίτερα στην υγεία και στις πιο ευάλωτες ε, ομάδες, τους νέους. Έχουμε πολλές προκλήσεις λοιπόν στις χώρες αυτές. Πρέπει να δούμε πώς συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, βιώσιμη ανάπτυξη με συμμετοχή όλων. Είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η ανάπτυξη αυτή βοηθήσει και την απασχόληση. Δουλειά για όλους. Και τους φτωχού και όσους βρίσκονται στο περιθώριο. Για τις χώρες ανατολικής γειτονίας τα προβλήματα αυτά έχουν μεγενθεί πολύ εξαιτίας της αύξησης των τιμών των αγαθών και της πολιτικής της Ρωσίας. Η Ουκρανία πλήττεται από μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση, για παράδειγμα. Η ελευθέρωση του εμπορίου με επενδύσεις θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε στις χώρες Ανατολικής Γετωνίας τα πλεονεκτήματα των στενών τους σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ συνεργαζόμαστε σε μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά προγράμματα τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Λευκορωσία. Συμμετέχουν εκεί οι πολίτες στο σχεδιασμό και στηρίζουν και την εφαρμογή κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή η κοινοτική για προγράμματα και στην ε, Ουκρανία ισχύει σε πολλές ε, περιοχές της χώρας, μετέχουν 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην περιοχή Ατζάρα τώρα, της Γεωργίας. Ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούν τους μικρούς αγρότες και τις, ε, τους του τους αγροτικούς. Στη Μολδαβία τα κοινά μας προγράμματα προωθούν την βιοενέργεια και την βιομάζα ως πηγή θέρμανσης στις αγροτικές περιοχές. Είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τέτοια κλίμακα. Έχουμε δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, επιχειρήσεις και βιομηχανίες εποφελούμαστε από την πρωτοβουλία More for More, περισσότερα και περισσότερα. Μια δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η περιοχή γεωπολιτικά είναι περισσότερο φορτισμένη μετά την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία. Που έχουμε επίσης και τις παγωμένες συγκρούσεις στην Απχαζία, Νοτιοσετία κλπ. κλπ. Ο ΙΕ προσπαθεί με δεύτερο τρόπο να βοηθήσει την Απχαζία και την Υπερδνηστερία παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εκεί επικεντρώμενοι στην βελτίωση της ζωής των κοινών ανθρώπων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων δίνοντας ε, χρήματα για τοπικές για παράδειγμα πρωτοβουλίες. Είναι πρωτοβουλίες από άνθρωπο σε άνθρωπο που χτίζουν την εμπιστοσύνη γιατί βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Στην Αρμενία Έχουμε επίσης μια επιτυχή πρωτοβουλία όπου βοηθάμε γυναίκες στην τοπική διοίκηση και τις προετοιμάζουμε να μπορούν να εκλογούν ώστε να συμμετέχουν περισσότερο οι γυναίκες στην πολιτική ζωή. Η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει ακρογωνίο λίθο της ε, πολιτικής της κυβέρνησης, τοπικά και περιφερειακά. Μια τρίτη πρόκληση έχει να κάνει με την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Επειδή είχαμε αυτήν την μια αποτελεσματική γραφειοκρατία και διαφορά την σοβιετική εποχή και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και αλλού, φαίνεται ότι μπορούν να γίνουν πράγματα. Οι χώρες αυτές πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό που εκείνες θέλουν και στο όραμα που έχουν και έτσι να χτίσουν μια στρατηγική πρέπει να δούνε οι ίδιες τι χώρα θέλουν να γίνουν και τι μέλλον θέλουν για τον εαυτό τους. Άρα διαφοροποίηση, ενστερνισμός είναι σημαντικά στοιχεία. Και ενώ η οικοδόμηση θεσμών είναι κάτι σημαντικό, πιο πολύ μας ενδιαφέρει η ποιότητα παρά η ποσότητα. Πώς μπορούμε να χτίσουμε και να ενισχύσουμε ε, την λογοδοσία, τη διαφάνεια υπέρ των ανθρώπων. Η σχέση μεταξύ των πολιτών και του κράτους επίσης είναι κάτι που δεν πρέπει να είναι θέμα ισχύω, πρέπει να είναι θέμα ε, σχέσης εκλογικής. Εταιρική σχέση τώρα ανάμεσα στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να βελτιωθεί η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Τα αποτελέσματα του ΟΗΕ είναι επιτόπου και προβάλλεται και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ παραλίλου και περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Συντονίζουμε επίσης τις δραστηριότητες του ΟΗΕ σε κάθε χώρο που έχουμε πρόσωπο. Επιπλέον, για την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη φέρουμε σε επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων, των ανθρώπων και έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έτσι μπορεί να υπάρχει μια καλή ανατολική γειτονία. Οι ωφελούμενοι λοιπόν έτσι βλέπουν καλύτερα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτούς. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να πετύχουμε τα ίδια πράγματα βάσει οικουμενικών αξιών και βάσει αυτού ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε μεταρρυθμίσεις και να βοηθήσουμε τις χώρες να πετύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Όλοι θα γνωρίζετε βέβαια τους στόχους της χιλιετίας. Το Σεπτέμβριο θα γίνει ο απολογισμό. Οι ηγέτες θα εγκρίνουν τη διώσιμη ανάπτυξη που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ατζέντα μας μετά το 2015, οι αξίες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντικατοπτρίζονται σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσοχή σας και περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σουλτάνογλου. Τώρα, περνάμε στους συντονιστές του ΟΗΕ. Ε, περαστικά στον κύριο Σαμαρασίνχα. Ελπίζουμε να τον δούμε κάποια άλλη στιγμή. Τρία λεπτά ο καθένας λοιπόν. Ξέρω ότι είναι λίγο, αλλά επειδή έχουμε πολλά θέματα και σας δω εκ των προτέρων συγγνώμη. Ο κύριος Βόκερ έχει τώρα Ουκρανία. αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, σας ευχαριστώ που φαίνεται τους επιτόπους συντονιστές των Ενωμένων Εθνών να σας μιλήσουν για τις ανατολικές χώρες μαζί σας, καθώς και την εργασία μας. Η εξέγερση του Μαϊντάν στην Ουκρανία έγινε κυρίως για ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για μια υπόλογη διάφανη κυβέρνηση, ένα τέλος στην διαφθορά, για να υλοποιηθεί η υπόσχεση του Μαϊντάν, η κυβέρνηση πρέπει να βρει βιώσιμη λύση στην σύγκρουση, να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Έχουμε 600.000 πρόσφυγες, 1,3 εσωτερικά εκτοπισμένους μέσα στην ίδια την Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης. Και πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέψουν σε εργασία. Early recovery το λέμε εμείς αυτό. Και χρειάζεται να γίνει και συστημική αλλαγή όλης της κυβέρνησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της κρίσης, ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του. Εργαζόμαστε εκεί για ανθρώπινα δικαιώματα, για την early recovery, για τις μεταρρυθμίσεις καθώς και για την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Εργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους εταίρους για να πετύχουμε γρήγορα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική στήριξη λαμβάνουμε σημαντική ενίσχυση από το πρόγραμμα ECO και ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή. Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερο φως για τα θέματα της early recovery και της μεταρρύθμισης. Τα προβλήματα αυτά της ε, έγκαιρης αποκατάστασης, της early recovery, δηλαδή να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους. Αυτό έχει ε, μεγάλη σημασία κάνουμε μια πρόταση 1,5 δισεκατομμυρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή είναι η λύση. Ακόμα περισσότερο και από την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις, συνταγματική, κοινοβουλευτική, κράτος δικαίου. Συνεργαζόμαστε στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, community development. Προωθούμε ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα ανάπτυξης των κοινοτήτων. Μπαίνουμε στην τρίτη φάση τώρα 2.500 κοινότητε σε όλη την Ουκρανία που μαθαίνουν πώ να κινητοποιούνται, πώ να κινητοποιούν του πόρου του για να επιτύχουν τι δικέ του προτεραιότητε στην καλύτερη διακυβέρνηση σε όλου του τομεί κοινωνικών κτλ. μέχρι και το περιβάλλον. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να συνεχίσει την σε βάθο στήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία και προσφέρουμε και τη συνεργασία με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών που διαθέτει και τεχνογνωσία και ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας δώσετε τόσες πληροφορίες σε τόσο λίγο χρόνο. Η κυρία Γαρτζέβα τώρα, Μολδαβία. Uh, Διακεκριμένε Πρόεδρε, ερήτημα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και ευχαριστώ που δίνετε δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες για την Μολδαβία όπου εκεί εργαζόμαι. Είναι πολλές οι συνιστώσεις και οι δυναμικές στη Μολδαβία. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση. Διαπραγματεύθηκε τη Συμφωνία Σύνδεσης επιτυχώς και την ε, πέρσι τον Ιούλιο και είναι η μόνη χώρα που μέχρι τώρα έχει ωφεληθεί από αυτή την υλοποίηση του τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική κρίση. Οφείλεται σε εξωτερικές και εσωτερικές εξελίξεις αυτό το γεγονός. Υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια και έχουμε και τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Έχουμε και οικονομική ύφεση στη Ρωσία, επιβράδυνση μάλλον, και έτσι εμβάσματα λιγότερα έρχονται και έχουμε και κλονισμούς στον φάτο εμπόριο. Αυτό έπληξε τον κοινωνικο ιστό της χώρας. Αντιμετωπίζει η χώρα πολλές προκλήσεις. Διαφθορά, τραπεζική κρίση, έλλειψη επιχειρηματικού κλίματος, προβλήματα δημογραφικά όπως διαρροή εγκεφάλων, μετανάστευση, γύρανση του πληθυσμού. Έχουμε και την παγωμένη σύραξη στην υπερνηστερία και ε, υπάρχει και έλλειψη ταυτότητας στον σοφατό Πρέπει να αντιστραφούν οι αρνητικές τάσεις. Χρειάζεται συγκροτημένη προσπάθεια από όλου του εταίρου αναπτυξιακού στη Μολδαβία, το πρόγραμμα του ΟΗΕ, το αναπτυξιακό, με συνεργασία άλλων φορέων του ΟΗΕ, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να στηρίξει τη χώρα, να στερνιστεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα μπορεί να καλύψει και τις αναπτυξιακές τη ανάγκες, τι βασικές. Έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση εδώ και χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τονίσω κάποια βασικά προγράμματα που έχουμε προγραμματίσει για να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες τις θεσμικές και να στηρίζουμε την τοπική κοινωνία, να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνη, να βελτιώσουμε τη ζωή του ντόπιου πληθυσμού. Έχουμε δύο προγράμματα. Μέτρα για ανάπτυξη εμπιστοσύνη, δημιουργία εμπιστοσύνη. Ενέργεια, βιομάζα. Μέσω των προγραμμάτων έχουμε βελτιώσει τη ζωή πάνω από 500.000 ανθρώπων. Έχουμε δημιουργήσει πολλέ θέσει εργασία. Και έχουμε εφαρμόσει και διασυνοριακά προγράμματα κατά τις δύο όχθες του Δνίστερου και θέλουμε να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέποντας όλα τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα με αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέρκεβα. Ο συντονιστής της Γεωργίας τώρα, ο κύριος Σκότ. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Θα εστιαστώ στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΟΗΕ στην αντιμετώπιση των κινδύνων από τι καταστροφέ, κυρίω ε, μετά σοβαρέ πλημμύρε που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη Γεωργία. Και να επαναλάβω τα συλληπιτήριά μου προ τι οικογένειε των θυμάτων. Τα τραγικά γεγονότα τόνισαν εκ νέου το βασικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων εταίρων συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ όσον αφορά τη στήριξη βιωσιμής και ισορροπημένης ανάπτυξη. σε συνθήκες που αλλάζουν γρήγορα στις χώρες αυτές. Δεν παρηγορεί αυτό τα οικογένειε των θυμάτων βέβαια. Τονίζουμε όμως ότι είναι σημαντική η ισορροπημένη πολιτική αντιμετώπιση των πλημμυρών. Επεξεργαζόμαστε μέσω των αναπτυξιακού προγράμματο του ΙΕ τα μέτρα αυτά. Απαιτεί τη δημιουργία υποδομών, δρόμων και άλλων υποδομών που διασχίζουν τις παιδιάδες που πλημμυρίζουν και μειώνουν την εισρωή των υδάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν συνηθισμένε πρακτικέ για τη μετώπιση των προβλημάτων αυτών. Χρειάζεται ορθολογική προσέγγιση όσον αφορά τη μετώπιση και τη δημιουργία λεκανών απορροής των υδάτων. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία υποδομών και της κυβερνήσεις να υλοποιήσουν αυτές οι υποδομές και να αναπτυχθούν σωστά. Τα γεγονότα στη Γεωργία μας υπενθύμισαν εκ νέου ότι οι φυσικές καταστροφές και οι συγκρούσεις μπορούν να εξαλείψουν ε, σε δευτερόλεπτα τα κέρδη της που αποφέρει η ανάπτυξη και μας υπενθυμίζουν αυτά με θλιβερό τρόπο ότι πρέπει να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο και μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ενθαρρύνοντας ισορροπημένη προσέγγιση για την μετώπιση των καταστροφών και την μείωση των σχετικών κινδύνων. Και μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΟΗΕ και άλλων εταίρων να προωθήσουμε την αποφυγή συγκρούσεων, την λύση των προβλημάτων και την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκότ. Ο κύριος Κουσέτα έχει το λόγο συντονιστής για την Αρμενία. Καλή σας μέρα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και εσείς αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε σήμερα για την Αρμενία και το όσα κάνει η οργάνωσή μας εκεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική χώρα στην περιφέρεια αυτή, κλειστή γύρω-γύρω, βέβαια πρόκειται για παγωμένη σύγκρουση και αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές και δημογραφικές προκλήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικό εταίρος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών στην Αρμενία και έχουμε κοινέ αξίες. Εργαζόμαστε μαζί σε πολλούς τομείς για να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα υπέρ του λαού της Αρμενία. Η έλλειψη ισότητα των φύλων παραμένει ένα σημαντικό θέμα στην Αρμενία δεν είναι μόνο πολιτικό θέμα η ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι και απώλειας οικονομικού δυναμικού. Πέρασε ένα σημαντικό νομοσχέδιο που καθιερώνει την ισότητα των δύο φύλων, αλλά φάνηκε ότι δεν είναι επαρκές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο UNDP εργάζονται για την συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε όλες τις, ε, ε, σε όλα τα επίπεδα της διοικήσεως και έχουμε μέχρι τώρα δείξει επιτυχία. Έχουμε χιλιάδες γυναίκες που έχουν διοριστεί σε θέσεις και έχουν εκλεγεί και πάνω από 60% των γυναικών που έχουμε εκπαιδεύσει εμείς. Αλλάζει σιγά σιγά η κοινωνία εφόσον αυτό επιτύχει σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερο, ένα άλλο σημαντικό, μια άλλη σημαντική πρόκληση, πώς να βοηθήσουμε την Αρμενία να βελτιώσει την διασύνδεσή της με το υπόλοιπο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται, της περιοχή στην οποία βρίσκεται και με τον υπόλοιπο κόσμο. Από το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το UNDP συνεργάζονται για να βελτιώσουμε τις διασυνδέσεις με την γεωργία, όχι μόνο με νέες υποδομές, αλλά και τη βελτίωση της κινητικότητας ανθρώπων και εμπορευμάτων και τη βελτίωση του εμπορίου που για τους ε, Αρμενίους αυτό το σύνορο είναι το πιο σημαντικό. Δεν μιλούμε μόνο για την ασφάλεια αλλά και για την ανάπτυξη για να συμπληρώσω την ε, σύντομη παρέμβασή μου, δεν πρέπει τώρα να αποσυρθείτε από την Αρμενία. Μάλλον να εμπλακείτε ακόμα περισσότερο στην Αρμενία μέσω της ε, πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξασφαλίσετε ότι θα διασυνδεθεί ακόμα καλύτερα με την μεγάλη οικογένεια όλων των εθνών για να μπορέσει να αναπτυχθεί την οικονομία της και την κοινωνία της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για το Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Αντώνιος Κρόινκ. Thank uh, Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Το Αζερμπαϊτζάν αυτή τη στιγμή ε, έχει υποδεχθεί τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες με θαυμάσιο τρόπο πραγματικά. Ε, μειώνονται βέβαια οι τιμές του πετρελαίου και αντιμετωπίζει προκλήσεις και η οικονομία τους όπως είπε και ο συνάδελφός μου εδώ δίπλα μου, παραμένει και η παγωμένη σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Στα θέματα της κυβερνήσεως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ένας τομέας όπου τα πηγαίνει πολύ καλά είναι η παροχή δημοσίων υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών βασισμένη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει δημιουργηθεί κέντρο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό η οργάνωσή μας, η UNDP, συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξετάζει και ελπίζω ότι θα εμπλακεί ακόμα περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ομάδες, νέοι, γυναίκες και άνθρωποι με αναπηρίες, πάλι εκεί η UNDP ε, εργάζεται για να προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης στις ομάδες αυτές και αντιλαμβανόμεθα ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει ιδιαίτερα στην επαγγελματική κατάρτιση προς όφελος των ομάδων που ανέφερα. Η οργάνωση UNDP αλλά και οι προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένους κέριους τομείς, για παράδειγμα στην βιώσιμη και ε, οικονομική ανάπτυξη για όλους στην διαχείριση του περιβάλλοντος και στην ανθεκτικότητα. Ιδίως δε σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης της υπαίθρου όπου υπάρχει σημαντική διασύνδεση των προτεραιοτήτων αυτών. Συνεργαζόμαστε θαυμάσια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησα και για ορισμένα από τα προγράμματά μας, Ένα, μια προσέγγιση βασισμένη στα οικοσυστήματα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Το Αζερμπαϊτζάν αντιμετωπίζει σοβαρές ε, ε, επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος με επιπτώσεις και στις τοπικές ε, κοινότητες που είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα. Ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε είναι η δουλειά που κάνουμε με την Civil Service Committee της οποίας ηγείται ο ίδιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την εφαρμογή του σχεδίου μεταρρύθμισης των θεσμών και έχουμε και ένα πρόγραμμα δημιουργία θεσμών και μια θαυμάσια συνεργασία μεταξύ Αζερβαϊτζάν, UNDP, Ευρωπαϊκής Ενώσεω και και συνολικά λοιπόν η συνεργασία μας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην οργάνωσή μας, η UNDP, είναι θαυμάσια και ε, στοχεύει σε ορισμένες εθνικές προτεραιότητες. Κάπου θέλουμε, όπου θέλουμε να εργαστούμε ακόμη περισσότερο είναι όχι μόνο η ποιότητα των παρεχόμενων, όχι μόνο η ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίω προ τι ευάλωτε ομάδε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σουτανόγλου και τη συγχαίρω για τους διακεκριμένους που έχει στην ομάδα της. Μπράβο τηρήσατε την πειθαρχία. Εμείς οι ευρωβουλευτές δεν τηρούμε τόσο πολύ, δεν πειθαρχούμε τόσο πολύ. Λοιπόν, συζήτηση τώρα. Οι ευρωβουλευτές παρακαλώ να ρωτήσουν αυτόν που θέλουν να ρωτήσουν, να πούνε ποιος είναι και όχι πάνω από τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πρέντα. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι χαίρομαι πολύ που σήμερα στην Επιτροπή μας έχουμε τους ε, επιτόπους συντονιστές των Ηνωμένων Εθνών για τις πέντε χώρες της Ανατολικής γειτονίας. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ο έκτος ήταν αδιάθετος και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας με τους συντονιστές αυτούς, διότι όπως έχει ήδη υποθεί πρέπει να υπάρχει συνοχή στη δράση μας. Έχουμε κοινούς στόχους μεταξύ μας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΙΕ, όσον αφορά την ευημερία, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την πολιτική λειτουργία των χωρών αυτών. Πρόσφατα συζητήσαμε μια έκθεση από αυτού για τις χώρες ανατολικής γειτονίας και έτσι, πράγματι, πρέπει να στηρίζουμε προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς, καλύτερη λειτουργία και διαφάνεια στους θεσμούς των χωρών αυτών, τήρηση κράτους δικαίου, συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή και βέβαια πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεπώς, θα ήθελα να γνωρίζω για το Αζερβαϊτζάν, επειδή να, ακούσαμε μόλις το συντονιστή στη χώρα αυτή, που είπε ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ίσως αθλητικά, πολιτικά όμως, η αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες εξαιρέσεις. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ο Ρουμάνος ήταν εκεί. Κατά τα άλλα όμως δεν πήγαν, πώς να το πω, πολιτικά. Δεν στηρίχτηκαν, ε, δεν στηρίχτηκε το πρωτάθλημα αυτό από πλευρά τη Ευρώπη. Ο ίδιο ο Τούρκο Πρωθυπουργό είπε γιατί λέμε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά παιχνίδια αφού δεν ήρθε κανένα Ευρωπαίο ηγέτη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συγγνώμη. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση ακριβώς με το πρωτάθλημα αυτό στο Μπακού, με ψήφισμα. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις για την κυρία Κερκεβά που είναι στην Μολδαβία για την ε, τρανσδιστερία και το σχετικό πρόγραμμα. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και υπάρχει κάποια δράση που να ασχολείται και με τους ρουμανόφωνους στην υπεδνηστερία. Όταν ήμασταν εκεί δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για τις εκλογές, για την παρατήρηση των εκλογών για παράδειγμα. Ήταν αδύνατον να τα καταφέρουμε. Οι Ρώσοι παραστρατιωτικοί μας εμπόδισαν. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω η χρηματοδότησή σας που πηγαίνει στην υπευνηστερία ποια είναι σε σχέση με το υπόλοιπο για τη Μολδαβία. Τώρα στον κύριο Βόκερ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι υπήρχαν παλιότερα πολλά προγράμματα στην Κρυμαία και στις περιοχές που σήμερα λέγονται αποσχιστικές. Έχετε προγράμματα που συνεχίζονται εκεί. Και ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις και το θέλει. Γιατί είπατε ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά στην Κρυμαία ο κόσμος μεταρρυθμίσεις περιμένει. Αυτό είναι το πρόβλημα, οι μεταρρυθμίσεις ή είναι η κατοχή. Οι άνθρωποι που είναι εκεί περιμένουν πράγματι μεταρρυθμίσεις, οι αποσχιστές, αυτοί τον πόλεμο θέλουν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μεταρρυθμίσεις εν καιρό πολέμου. Αυτή είναι η κατοχη οι ανθρωποι που ειναι εκει περιμενουν πραγματι μεταρρυθμισεις οι αποσχιστέ, αυτοι τον πολεμο θελουν μπορουμε λοιπον να κανουμε μεταρρυθμισεις εν καιρο πολεμου αυτη ειναι η ερωτηση μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέτα. Ο κύριος Πλίνκοβιτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, χαιρετίζω την κυρία Σουτάνογλου ξανά στην Επιτροπή μας και όλους εκπροσώπους των υπηρεσιών του ΟΗΕ στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Εκτιμώ τα όσα μας είπατε και τη συνεργασία μας που είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της UDNP. Είναι πολύ χρήσιμη η παγκόσμια παρουσία σας Πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχόλιο για την κυρία Σουλτάνογλου. Μία ερώτηση ίσως για να κατανοήσουμε ποιος είναι ο προπολογισμό των φορέων του ΟΗΕ στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Να καταλάβουμε η ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική ένταξη, η ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων κλπ. Πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι προσπάθειες. Και πώς είναι η συνεργασία στο τοπικό επίπεδο με τον ΟΗΕ, πώς γίνεται η απορρόφηση των πόρων. Σαν Κροάτης εκτιμώ το ρόλο του ΟΗΕ, μας βοήθησε εδώ και 17 χρόνια να εφαρμόσουμε την ενόμη τάξη στη χώρα μου. Και εργάζεσαι σε χώρες όπου δεν είναι εξασφαλισμένη η δαφική ακαιρεότητα. Έχουμε και την πρόσφατη έκθεσή μας για την πολιτική γειτονία και έχουμε πολύ καλά παραδείγματα. Η μόνη επιτυχέστατη αποστολή του ΟΗΕ ήταν η μεταβατική διοίκηση της Ανατολικής Σλοβενίας στηρίχθηκαν οι εταίροι, απεκαταστάθηκε η πολιτική ε, αξιοπιστία και απεκαταστάθηκε η ακεραιότητα της χώρας μου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχετε υπόψη σας πάντα, είτε αφορά τη Μολδαβία, τη Γεωργία, είτε την Ουκρανία. Έχετε αυτή την εμπειρία, μπορείτε να βασιστείτε πάνω σε αυτή και μπορείτε να ε, προωθήσετε τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίτκινς έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω λετωνικά, λέει ο κ. Μάμκινς. Έχω μια ερώτηση για τον συντονιστή της Λευκορωσίας. Είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας συνεργασίας με τη Λευκορωσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή την εβδομάδα θα γίνει επίσκεψη στη Λευκορωσία. Ερώτηση τι αλλαγές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη Λευκορωσία εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Αισθάνεστε ότι ο εκδημοκρατισμός προωθείται όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης ή της ΜΚΟ. Αισθάνεστε να πνέει άνεμος αλλαγή στη Λευκορωσία. Ευχαριστώ. Εγώ εκ μέρου τη ΚΟΕ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βόκερ. Έχουμε διαφορετικέ απόψει, ίσω δικιά μα να μην είναι η πλειοψηφική, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να πούμε ότι εκείνοι που μετατοπίζονται εσωτερικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω ότι ο ΙΕ προσπαθεί να βοηθήσει, αλλά η ακραδεξιά, ασόφ και έχει προγράμματα για να στηρίξει τη δραστηριότητά σα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοχμπίλερ. Η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους σας. Θέλω να ρωτήσω για τις παγωμένες συγκρούσεις. Κυρίως τον εκπρόσωπο για την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Είπατε ότι έχετε εκεί κάποια προγράμματα. Έχετε και διασυνοριακά προγράμματα με συνεργασία μεταξύ σας. Και όσον αφορά τη Γεωργία, θέλω να ξέρω, υπάρχουν Γεωργοί που ζουν από τη μια μεριά της διοικητικής γραμμής, την Επχασία και την ε, Νότιο Σετία, αλλά η γη τους που καλλιεργούν βρίσκεται από την άλλη μεριά της διοικητικής αυτής γραμμής. Και έπειτα, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, το έθεσε και ο κύριος Πρέντα για το Αζερβαϊτζάν. Θέλω και εγώ να προσθέσω, γιατί είπατε ότι το πρωτάθλημα είναι επιτυχές. Ναι, είναι επιτυχές, γιατί δείχνει την κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν κάτω από τους προβολείς της επιτυχίας. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ανάλυση το πρωτάθλημα αυτό μάλλον οδήγησε σε περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, οι δημοσιογράφοι, οι ντόπιοι αλλά και ξένοι εμποδίστηκαν να παρουσιάζουν την κατασκευή. Υπάρχουν και πολιτικοί κρατούμενοι. Οπότε, καλό θα ήταν να ακούσουμε και από εσά, εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση. Υπάρχει βελτίωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριο Σκούκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ειλικρινά καλώς ε, ήρθατε, θέλω να πω και στην κυρία Ζουλτάνογλου και σε όλους τους επιτόπους συντονιστές του ΟΗΕ στις ε, χώρες Ανατολικής Γειτονίας. Έρχεστε μια πολύ σωστή στιγμή εδώ, μια από την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε την έκθεση όσον αφορά το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανατολική Γειτονία και εγώ ήμουν εισηγητής. Οπότε πολύ χαίρομαι που μπορώ να συζητήσω μαζί σας και θέλω να σας ρωτήσω για τη δυναμική που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αναπτυξιακά προγράμματα του ΟΙΕ. Υπάρχει εταιρική σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κύριος δωρητής Ποια, πώς πάει η συνεργασία με τον ΟΗΕ και πού θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή. Επίσης, πώς επικοινωνούμε τις προσπάθειές μας προς τον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε όταν προετοίμαζα την έκθεσή μου, το θέμα της προβολής μας, πώς προβάλλουμε το έργο μας. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε, να δείξουμε τι κάνουμε, ώστε ο κόσμος στις χώρες αυτές να καταλάβουν καλύτερα τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο χρήσιμη τους είναι δεν συμφώνησαν όλοι, οπότε πολύ θα ήθελα να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, Απχασία, Σετία, Υπερδνηστερία, πού είναι οι κύριες διαφορές και πού ο ΙΕ τα καταφέρνει καλύτερα. Δεν μίλησα ούτε δύο λεπτά, Πρόεδρε ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάρμπερ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μοναδική θέση του Αζερβαϊτζάν όσον αφορά τις ειδικές σχέσεις με το Ισραήλ. Είναι δίπλα στο Ιράν, χώρα με και επηρεάζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ποια είναι η υποψή σας? όσον αφορά τη θέση του Αζερβαϊτζάν στα πλαίσια της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν το γύρο των ρωτήσεων, ο κύριος Πέτερ λέει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα εισαγωγικά σας λόγια και για τη δουλειά που κάνετε στην περιοχή. Χαίρομαι που τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στενά, διότι βέβαια όλοι εργαζόμεθα επί βάσης κοινής, επί των ιδίων αξιών και μπορούμε μέσα της συνεργασίας να πετύχουμε τη θέμενη αξία. Όμως η περιοχή αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις Υπάρχουν πολλά απρόβλεπτα γεγονότα που καταφθάνουν πιθανότατα, οπότε βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η καλύτερη διακυβέρνηση. Χωρίς καλή διακυβέρνηση οι μεταρρυθμίσεις θα είναι ανεπιτυχείς. Υπάρχει κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερος, ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της ε, χρηστής διακυβέρνησης. Τι έχετε αποκομίσει από την εμπειρία σας. Λοιπόν, για να κερδίσουμε χρόνο. Προτείνω να αρχίσουν με την απάντηση οι συντονιστές με την ίδια σειρά και στο τέλος θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουλτάνογλου. Ο κύριος Μάμικιντς κάτι ρώτησε για τη Λευκορωσία, οπότε ίσως εσείς θα μπορούσατε να απαντήσετε γι' αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ. Ετέθησαν μία-δύο ερωτήσεις που με αφορούσαν. Το η πρώτη αφορούσε την Κρυμαία. Είναι σημαντικό να ξεκινήσω τονίζοντας ότι η Γενική Συνέλευση του ΕΕ ψήφισε ένα ψήφισμα που σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα της Κρυμαίας πριν από την κρίση. Τι σημαίνει αυτό. Ότι η Κρυμαία είναι κατεχόμενη περιοχή σύμφωνα με το ψήφισμα. Ο δεν είναι πρόσδεκτος στην Κρυμαία. Δεν είναι αποδεκτό ούτε από την κυβέρνηση Ουκρανίας ούτε τη Ρωσία. Υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι γι' αυτό. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε. Μπορώ, αν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βασικά δεν εργαζόμεθα εκεί τώρα. Έχουμε όμω το ψήφισμα που σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα τη Κρυμαίας. Είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ των εδαφών που κρατούνται από μη κυβερνητικού φορεί στην περιοχή του Ντομπά. Αυτέ οι περιοχέ καλύπτονται από τις συμφωνίες τις συνευτικές του Μίνσκ και πρόκειται να επανενταχθούν στην Ουκρανία και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία θέλει κάτι διαφορετικό, ενθαρρύνουν τους αποσχιστές ε, να βρουν μια λύση για μια ενιαία Ουκρανία. Η κατάσταση λοιπόν στην Ουκρανία και στο Ανατολικό Ντομπάς είναι διαφορετικές. Τώρα μεταρρύθμιση και εργασία μπορεί να και τα δύο η κυβέρνηση στην Ουκρανία πρέπει να ασχοληθεί με θέματα ασφαλείας και σύγκρουσης, με ανθρωπιστική κρίση και να αντιμετωπίσει τη μεταρρύθμιση. Πιστεύω ότι ειλικρινά θα πρέπει να τα καλύψει όλα. Δεν έχει επιλογή η κυβέρνηση. Είναι τεράστια πρόκληση. Θα ήταν τεράστια πρόκληση εδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και γι' αυτό η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρισίμου σημασία. Όπω τα βλέπω εγώ τα πράγματα, εργάζονται και επί των τριών τομέων. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, έχουν πολλά προβλήματα. σε λεπτομέρειε. Ουσιαστικά όμω ο πρόεδρο Μποροσέγκο ε, έχει σαφείς δεσμεύσεις και για τους τρεις τομείς. Υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη εντός της Ουκρανίας ε, που στηρίζει τη δράση και στα τρία μέτωπα και υπάρχει και στήριξη από τη διεθνή κοινότητα την οποία ανεκτιμούν πολύ. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τους εσωτερικά εκτοπιστέντες. Πρέπει να βρούμε πολύ δύσκολη ισορροπία εδώ, δηλαδή να ανταποκριθούμε σε απαιτήσει ανθρωπιστικές όσοι φύστανται, αλλά να κινηθούμε τάχιστα προς ε, έγκαιρη ανάκαμψη ε, στέγαση, εργασίες, να επενδύσουμε στα κοινοτικά κέντρα, στους χώρους που πρέπει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκε με την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΗΕ για να παράξει ένα πρόγραμμα ε, γρήγορη ανάκαμψη και αυτή είναι η πραγματική ανταπόκριση που χρειάζεται. Εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι το εξή, ότι η αναπτυξιακή πτυχή τη ταχεία αναπτύξεω είναι πιο αργή να ξεκινήσει από ό,τι ανθρωπιστική πτυχή και δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα να δίνουμε μια συνέχεια όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια μακροχρονίως όταν η απάντηση είναι η ανάπτυξη. Και στα 7 δευτερόλεπτα που απομένουν θέλω να πω ότι το δεύτερο τμήμα της ερωτήσεως αφορούσε την πολιτική σταθερότητα, αν το ερμηνεύω σωστά. Θέλω να πω ότι η συμμαχία, ο συνασπισμός στην Ουκρανία, η συμμαχία στην Ουκρανία είναι πολύ εύθραυστη. Είναι κατανοητό αυτό, έχει μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει κρίση. Ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός ε, ανέλαβαν την υποχρέωση να εργαστούν και είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ότι ε, θα εξακολουθεί να, να κρατάει ο συνασπισμός αυτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσον αφορά τη Μολδαβία, λέει και η Γκέρκεφα. Πρώτα απ' όλα για την υπερδυνστερία. Πράγματι στην υπερδυνστερία... Η UNDP είναι από τους λίγους εταίρους στους αναπτυξιακούς που έχει πρόσβαση στην επικράτεια και είναι πρόσδεκτος από τις de facto αρχές. Εφαρμόζουμε δύο προγράμματα στην Περνιστερία που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τα μέτρα εμπιστοσύνη και ενέργεια και βιομάζα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι εδώ στο πλαισίου των δύο προγραμμάτων και των έργων έχουμε πολλά από τα αποτελέσματα που επέδευξαν και στην πρώτη φάση του προγράμματος οικοδόμηση εμπιστοσύνη. 13 νέες πρωτοβουλίες θα εφαρμοστούν 15, μάλλον 30, 15 από τη μία όχθη, 15 από την άλλη όχθη του Δνίστερου. Είναι πρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες από την τόπια κοινωνία και από τις αρχές και έχουμε πρόσβαση σε κάθε χωριό και κοινότητα όπου υπάρχουν ανάγκες και εντοπίζονται αυτές από τους τοπικούς δικαιούχους και συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε και ερώτηση όσον αφορά την ορατότητα και θέλω να πω ότι η ορατότητα είναι μια διαδικασία και όχι αυτοσκοπός, απαιτεί συνεχή εστιασμένη προσπάθεια. Είναι κάτι εξίσου σημαντικό και πιστεύω ότι καταφέραμε να πετύχουμε άριστα αποτελέσματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση των δικαιούχων από τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τους ενημερώνουμε περί της αξίας της αποδοχής αυτής της βοηθείας, και πώ ένα πλησίασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιώσει τι συνθήκε διαβίωσή του και θα του δώσει δυνατότητα για ανάπτυξη, ασφάλεια και ευημερία. Υπήρξε μια ερώτηση που αφορούσε τη χρηστή διακυβέρνηση και πώ μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω αυτή και να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί η δημοκρατία και ότι είναι αποτελεσματική η διακυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επιβληθεί έξωθεν, πρέπει να αναπτυχθεί έσωθεν. Και ένα κρίσιμο στοιχείο είναι να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχει η κοινωνία των πολιτών. Χωρί ισχυρή και βιώσιμη κοινωνία των πολιτών, πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Σκότ. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είχε να κάνει με τη διοικητική γραμμή την Γεωργία. Ρωτήσατε αν υπάρχουν ε, ενισχύσεις προς τους αγρότες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ελεύθερη κυκλοφορία κυρίως και όχι τόσο με την γεωργία αυτή καθεαυτή έχει να κάνει και με την υγεία και με την εκπαίδευση, με επισκέψεις στους συγγενείς τους, ε, σε τάφους των προγόνων τους κλπ. κλπ. Έχουμε μια πρόσφατη έκθεση του Προσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρεται στις προσβάσιμες περιοχές του κόσμου για την Νότια Οσετία. Και συνεχίζουμε να μελετάμε το θέμα και συνεχώς λέμε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να τηρούν τις συμφωνίες και να μην υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί. Όσον αφορά την βοήθεια, πάντως, ναι. Και εδώ θα περάσω στη δεύτερη ερώτηση που λέτε ποιες είναι οι επιτυχίες σας όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Εδώ θέλω να αναφερθώ σε ένα πρόγραμμα που ονομάζουμε COBAM και είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα που στηρίζεται συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία πέντε χρόνια και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και στην Απχαζία, την Ανατολική και τη Δυτική μεταξύ των κοινοτήτων που ζουν εκεί δηλαδή. Και έχει βοηθήσει και στο πρόβλημα Γεωργίας ε, Απχαζίας. Με συμμετοχή διάφορων μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων. Απχαζία, Νότιο Σετία κλπ. Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η συνεργασία εδώ στο πρόγραμμα αυτό, ο ΙΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα από τα λίγα διεθνή προγράμματα που στηρίζουν τη κοινωνία των πολιτών ε, και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Νότια Σετία. Υπάρχουν βέβαια επικρίσεις για κατασκοπίες κλπ. Είναι προβληματική προβολή του έργου μας στην ε, Νότια Σετία. στην Απχαζία όμως είναι θετική αξιολόγηση. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είναι ορατό το έργο μας. Τέλος για την χρηστή διακυβέρνηση, τρίτη ερώτηση που θα απαντήσω για τη Γεωργία. Πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης είναι, όπως είπα και νωρίτερα, ιδίως τώρα με τις πλημμύρες που προέκυψαν, κάτι στοιχειώδες. Αλλά έχει να κάνει και με την οικονομική ανάπτυξη. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική η οποία μακροπρόθεσμα να βοηθάει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώς, η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων όχι μόνο στην γεωργία, αλλά παντού θα βοηθήσει την πολιτική ανατολικής γειτονίας. Ευχαριστούμε. Επόμενος. Όσον αφορά τη δουλειά που κάνουμε, σε τομείς που υπάρχουν οι παγωμένες συγκρούσεις, ο ΙΕ στην Αρμενία δεν έχει εντολή να λειτουργήσει στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Στηρίζουμε την ομάδα του Μιν στο βαθμό που μπορούμε, αλλά δεν έχουμε δραστηριότητες στην επικράτεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ για τη χρηστή διακυβέρνηση. Βασικό ερώτημα. Για την Αρμενία. Και εκεί προσπαθούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταπολέμηση διαφθοράς και συμμετοχή των πολιτών. Το ανέφερα αυτό. Συνεργασία με, τους, ε, με τις γυναίκες και με τους ντόπιου πληθυσμού. Στην Αρμενία υπάρχουν προβλήματα. 1% του πληθυσμού με τα αναστεύει από τη χώρα κάθε, κάθε χρόνο. Βασική πρόκληση οι νέοι να παραμείνουν στη χώρα, να ασχολούνται με τα ζητήματά της και να καταπολεμήσουμε τη γενική απάθεια. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να διαμορφώσουμε συμμετοχική δημοκρατία. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει πρόγραμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύντομα με άμεση συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους επόμενους μήνες θα υλοποιηθεί. Θα καλύψουμε διάφορα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αρμενία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί αγώνες έχουν προσελκύσει πολύ προσοχή τώρα. Από πλευράς ΟΗΕ δεν είμαστε μέλος Είμαστε, είμαι εξωτερικός παρατηρητής. Πολύ προσοχή δίδεται στα, στους αγώνες. Υπάρχουν και πολλοί αθλητές από την Αρμενία που συμμετέχουν. Αυτό είναι θετικό, αξιέπαινη συνεργασία. Έχουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης. Ενεργοποιούμεθα σαν ΟΗΕ μαζί με διάφορους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την UNPR, την, ε, το, και θα συνεργαστούμε με τους φορείς για να στηρίξουμε τη χώρα, να υλοποιήσουμε τις συστάσεις που έχουν γίνει. Πριν από μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση πήγε στη Γενέβη και ο συνάδελφός μου και εγώ που ασχολούμεθα με τα γυναικεία δικαιώματα συμμετείχαμε στην αναθεώρηση του ΣΥΝΤΟ και θα δώσουμε συνέχεια σε όλα τα ζητήματα. Ασχολούμεθα με τα δικαιώματα των γυναικών, την έμφυλη βία, συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή την Αρμόδια για θέματα γυναικών, οικογενειών και παιδιών για τις παγωμένες συγκρούσεις. Δεν έχουμε εντολή, όπως προανεφέρθηκε γι' αυτό. Έχουμε προγράμματα όμως ταυτόχρονα με την Αρμενία, τη Γεωργία, το Ατζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία. Έμεσα τα προγράμματα αυτά ωφελούν τις χώρες και μπορούν να γίνουν περισσότερα Κάποιος αναφέρθηκε στο Ισραήλ. Δεν γνωρίζω πολλά από γεωπολιτικά ζητήματα. Ξέρω ότι όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και η εβραϊκή κοινότητα του Αζερμπαϊτζάν είναι σε πολύ καλή θέση. Η χώρα προωθεί την ανεξιθρησκεία και οι ομάδες οι εβραϊκές και άλλες θρησκευτικέ ομάδες και μειονότητες αισθάνονται αρκετά άνετα και το Αζερβαϊτζάν ε, δραστηριοποιείται διοργανώνοντας διεθνείς συναντήσεις που αφορούν την ανεξιθρησκεία και την ανοχή των διαφόρων πολιτισμών. Θα σταματήσω εδώ. Συνεργαζόμαστε στενά με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Αζερβαϊτζάν. Συζητούμε αυτά τα θέματα, πώς από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Αυτά και ευχαριστώ. Και ξεπέρασα τα τρία λεπτά μου. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω ποιος για τον κύριο Χάφικ, αν θα μιλήσει κάποιος πριν δώσω τον λόγο στην κυρία Σουτάνογλου. Όχι, κυρία Σουτάνογλου τότε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους αξιότιμους ευρωβουλευτές. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις και σημαντικό το ενδιαφέρον που δείχνεται για τις δραστηριότητές μας και στην κοινή μας συνεργασία την οποία χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες από τις πιο γενικές σας ερωτήσεις. Ασφαλώς οι εκπρόσωποι των χωρών δηλαδή οι εκπρόσωποι του στις χώρες. Σας έδωσα μια εικόνα του έργου μας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, παρακαλώ, ευχαρίστως να έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω του γραφείου συνδέσμου μας εδώ, η UNDP είναι και αρμόδια για τον ε, δίκτυο διαφάνειας. Κάθε πληροφορία που χρειάζεστε λοιπόν είναι διαθέσιμη εδώ. Τώρα για τη Λευκορωσία, ο συνάδελφός μας βέβαια λείπει σήμερα. Αυτό που βλέπουμε πράγματι και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσά θα συμφωνήσετε είναι μια, ένα σταδιακό άνοιγμα. Μια εκδήλωση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από την πλευρά της κυβέρνησης της χώρας αυτής να εμπλακούν σε αυτά που λέμε εκδημοκρατισμός, καλή διακυβέρνηση, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίσως τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να φύγουν πλέον από τον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και να πούν κάπου αλλού. Εμείς είμαστε βέβαια, στον, συμμετέχουμε στον διάλογο αυτό, δεν είναι διάλογος άλλωστε ο οποίος μόλις ξεκίνησε, έχουμε εργαστεί από καιρό για αυτόν και εν τέλει πρόκειται για μια διαδικασία συνεχιζόμενη δηλαδή θα γίνει δεν θα ολοκληρωθεί από τώρα μέχρι το φθινόπωρο. Είναι σωστό νομίζω να πούμε ωστόσο ότι πνέει ένα άνεμος αλλαγής. Η συναδελφό μα από την Αρμενία νομίζω είπε, ή από το Αζερβαϊτζάν δεν είμαι βέβαιος, είπε για, αυτήν, για αυτό το όργανο των Ηνωμένων Εθνών και την παρακολούθηση των εξελίξεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λευκορωσία Είχαμε την Διεθνή Σύμβαση για τα Δίκαια των Ανθρώπων με Αναπηρίες ως entry point. Και τώρα ε, μιλούμε για ένα είδος σχεδίου δράσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίζουμε επίσης και την κοινωνία των πολιτών για πολλά χρόνια είτε άμεσα είτε έμεσα με πολλά έργα που διεξάγονται στο τοπικό επίπεδο και project τα οποία γίνονται για ε, τον ιό του AIDS, για πρόσωπα που έχουν, ε, είναι φορείς ή έχουν ε, ασθενήσει από τον ιό του AIDS και αυτά βοηθούν για να αναπτυχθεί το θέμα. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Στα αρχικά στάδια έχουμε όμως την μεγάλη ελπίδα ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση και ποιες δυνατότητες έχουμε στην περιοχή αυτή. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τα Δυτικά Βαλκάνια, την Αλβανία, τον Κάφκασο και πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας και την Τουρκία και έχουμε και διακοινωτικές συνεργασίες στην Κύπρο με συνεργασία του Οργανισμού Ενωμένων Αθηνών και της Ένωσης. Είναι λοιπόν πολλές οι χώρες και δεν έχουμε τακτικούς πόρους που να δίνονται για τις χώρες αυτές. Άρα οφείλουμε να συνεργαζόμαστε σε στενή συνεργασία και με άλλους. Στην περιοχή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους μεγαλύτερους εταίρους μας. Μαζί με ορισμένες διμερείς προσπάθειες, όχι και τόσο διμερείς πάλι βέβαια για τους λόγους που εξήγησα πριν, και αυτό που αποκαλούμε ταμεία για ειδικού σκοπούς, περιβάλλον, HIV, AIDS κλπ. Όλο και περισσότερο βέβαια βασιζόμαστε στη συνεργασία των κυβερνήσεων. Γιατί οι εγχώροι πόροι είναι πολύ σημαντικότεροι και για την κυριότητα της ανάπτυξης, για την ownership δηλαδή. Συνεργαζόμαστε λοιπόν πολύ περισσότερο από πριν με τις ίδιες τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, έτσι ώστε να αφιερωθούν τμήματα του προϋπολογισμού στις δραστηριότητες που θέλουμε να προωθήσουμε. Πέρσι φτάσαμε σε συνολικό ποσό περίπου 370 εκατομμυρίων δολαρίων. Φέτο αναμένουμε να φτάσουμε περίπου τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μεγάλο μέρο, δηλαδή ένα τεράστιο μέρο από αυτά προέρχεται από εταιρικέ σχέσει που ανέφερα πριν, partnerships. Σε ό,τι αφορά την κατανομή, το συζητούσαμε αυτό εδώ με τον συναδελφό μου Γιάννη πριν από λίγο, είναι περίπου το 1 τρίτο. Αλλά δεν υπάρχουν εκεί τις διαχωριστικές γραμμές. Όσον αφορά τώρα την συνεργασία με τις κυβερνήσεις, μίλησα για την υπόθεση της Λευκορωσίας, αλλά και οι συνάδελφοί μου απείδησαν σχετικά. Όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και εμείς πολυετή προγράμματα, στη δική σας περίπτωση όχι για όλες τις χώρες, στη δική μας περίπτωση για όλες τις χώρες, εκτός από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, όλες οι χώρες στην ε, περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας έχουν νέα προγράμματα από το 2016 μέχρι το 2020 και εκεί προωθούμε τις προτεραιότητες που διαθέτουμε όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας ε, στις ε, χώρες αυτές. Έχουμε, μιλούμε για αηφόρο ανάπτυξη, κοινωνική συμπερίληψη, δουλειές, περιβάλλον και καλή διαχείριση, καλή διακυβέρνηση. Αυτά προσφέρουν ευκαιρίες και σε εμά να προωθήσουμε τα θέματα που μας απασχολούν για την ατζέντα μετά το 2015 βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των προσπαθειών μας. Κάναμε λοιπόν έρευνες στην περιοχή αυτή με πολύ καλή συμμετοχή, διαβουλεύσεις ε, με πανεπιστημιακούς, με την κοινωνία των πολιτών, με κυβερνήσεις, επίσης και online ζητώντα να μα πούν οι άνθρωποι τι αναμένουν για το μέλλον. Και ακούσαμε, ανεξαρτήτως χώρας, αυτό που ακούσαμε ήταν κυρίως τρία πράγματα, βέβαια με αλλαγή προτεραιότητε, προτεραιότητες, αλλά τα τρία ήταν πάντα τα ίδια. Δουλειέ, ποιοτικέ υπηρεσίες στέγη και παιδεία και έντιμη και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Αυτές είναι βασικά οι προτεραιότητες μας. συμπεριλαμβανομένης και της νέας πολιτικής για την ENP. Και η προσπάθειά μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να φτάσει στους στόχους αυτούς. Ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα ήδη, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους κύριους εταίρους μας και διαρκείας μάλιστα και παγκοσμίω, όχι μόνο στην περιοχή αυτή του κόσμου. Αυτό που μας απασχολεί τα τελευταία δύο χρόνια και που έχουμε στοχεύσει είναι να αναγάγουμε την εταιρική αυτή σχέση σε στρατηγική εταιρική σχέση. Όχι λοιπόν μόνο στο επίπεδο του συγκεκριμένου έργου, project level, αλλά και για το τι οφείλει να γίνει συνολικότερα. Αυτή λοιπόν η στρατηγική ε, εμπλοκή σημαίνει και στο τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο χώρας ότι τα γραφεία των χωρών συνεννοούνται με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για προγράμματα που αφορούν την ίδια τη χώρα είτε για διάφορα εργαλεία τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για προγραμματισμό και για υποβολή εκθέσεων, reporting. Γνωρίζουμε καλά το γεγονός ότι η εδίποτε εταιρική σχέση θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει προς τη θέμενη αξία. Γνωρίζουμε επίσης το ενδιαφέρον των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργαστούν πιο στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αυτό είναι κατανοητό. Εμείς τονίζουμε επίσης το γεγονός ότι είναι πολύ διαφορετικές οι πτυχές της εταιρικής αυτής σχέσης λόγω και των λόγων που ανέφερα στην αρχική μου τοποθέτηση, όχι μόνο λόγω ουδετερότητας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών βέβαια και της παγκόσμιας θέσης του, αλλά και των αξιών που είναι παγκόσμιες αξίες, ειρήνη, σταθερότητα, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αυτά λοιπόν είναι απλά πράγματα. Τώρα για την ορατότητα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ίσως να μην τα καταφέραμε τόσο καταπληκτικά στο παρελθόν για να υποστηρίξουμε αυτή την απέτηση ορατότητας που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα καταφέρνουμε τώρα καλύτερα και βλέπουμε και από τις πρόσφατες εμπλοκές που έχουμε ότι μπορέσαμε να προσφέρουμε μεγαλύτερη ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απόλυτα ότι η ορατότητα δεν σημαίνει μοναχά λάβαρα και πινακίδες, αλλά οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι να κατανοήσουν ότι αυτό που λαμβάνουν είναι μια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να επιτευχθούν θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Αυτή η ορατότητα λοιπόν θα πρέπει να είναι στην καρδιά κάθε προσπάθειας. Και οι δικαιούχοι οι άνθρωποι, οι πολίτες να κατανοήσουν ότι αυτά που λαμβάνουν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την προοπτική αυτή. Θα είναι σημαντικό νομίζω όσο προχωρούμε να δείξουμε κάποια ταχεία και κάποια ευκαμψία στην διαδικασία αξιολόγηση, διότι υπάρχουν τα διάφορα επίπεδα. Υπάρχει το επίπεδο της πολιτικής policy level, ε, της ε, λήψης αποφάσεων και τα καθεξής. Οι περισσότεροι όμως στα πιο χαμηλά επίπεδα δεν το κατανοούν αυτό. Πώς λοιπόν θα φτάσουμε μέχρι το επίπεδο αυτό και πώς θα τους προσφέρουμε τα απαραίτητα το δυνατόν συντομότερο. Βλέποντας και τις ικανότητες που έχουμε επιτόπου, ποιες είναι οι δυνατότητες δηλαδή να εφαρμόζουμε τα προγράμματα, μπορούμε να συνεχίσουμε μια κοινή προσπάθεια για να επιτύχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα υπέρ των ανθρώπων στο τοπικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν και εδώ ολοκληρώνω την παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και για την ποιότητα των παρουσιάσεών σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε ειλικρινά. Ήταν πολύ καλό που είχαμε αυτήν την συνάντηση. Και να ξέρετε, το λέω εγώ που προεδρεύω εδώ, ότι η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή για τα Ηνωμένα Ωραία. Περιμένουμε μέχρι 10.30 για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. no, no, no. Vamos a comenzar con el... Προχωράμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο μας. Καλωσορίζω λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά εδώ τον Φιλίπ Ντούστ Μπλαζή που είναι Γενικός Υπογραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Θα μας μιλήσει για τη χρηματοδότηση των προτεραιτήτων για την ανάπτυξη. Είναι και πρόεδρος της Unicite που είναι μια οργάνωση η οποία αγωνίζεται για καλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλίσουμε πρόσβαση σε θεραπείες και σε διάγνωση για το AIDS, την ολονοσία και τη θυματίωση στις πιο φτωχές χώρες. Όπως γνωρίζετε, εκτιμάμε όλος ιδιαίτερο τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί πιστεύουμε ότι η Ηνωμένα Έθνη είναι ένας εταίρος αναγκαίος για να φτάσουμε να βοηθήσουμε εκεί που θέλουμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τις προηγούμενες εβδομάδες ακούσαμε δύο σημαντικές προσωπικότητες των ΗΠΑ, τον που είναι ο Γενικός Γραμματέας, και τον κύριο Κουτέσα, που είναι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Και οι δύο λοιπόν υπογράμμισαν ότι χρειάζεται μια συνεργασία και μεγαλύτερη ακόμα για να αντιμετωπίσουμε τους στόχους μας και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλά. Το 2010 λοιπόν είναι μια καλή στιγμή για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι εσείς είσαστε από αυτούς που προωθούν ένα νέο και πιο φιλόδοξο πλαίσιο συνεργασίας. Όλοι μας, όλες οι χώρες πρέπει να αντιληφθούμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η μετανάστευση είναι αλληλένδετα και ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού απαιτούν ανάπτυξη πρώτα απ' όλα. Πρέπει να προβλέψουμε φιλόδοξα μέσα για την ε, εφαρμογή της ατζέντα μας για μετά το 2015. Οικονομικά μέσα πρώτα απ' όλα, επίβλεψη και υπευθυνότητα. Είσαστε εδώ για να μας ε, παρουσιάσετε τις θέσεις σας για αυτές τις κοινέ προτεραιότητες που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη για το μέλλον. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 10 λεπτά προκειμένου μετά να ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Με τιμάει. Ήμουνα Ευρωβουλευτής το 89 με το 93. Οπότε πρέπει να σας πω ότι σέβομαι πάρα πολύ το χώρο αυτό και το σώμα αυτό. Δέκα λεπτά μου δώσατε, είναι λίγα μεν, αρκετά όμως. Θα πω γρήγορα. Το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα ίσως είναι το θέμα υπαρτιμών ένα διεθνούς πολιτική στον κόσμο. Ο πρόεδρος Λούλα συνήθιζε να λέει όταν ήταν στην Προεδρία στη Βραζιλία ότι Δεν είναι στο Ιράν ή στη Βόρεια Κορέα που έχουμε το μεγαλύτερο ατομικό κίνδυνο. Ο μεγαλύτερος ατομικός κίνδυνος, πυρηνικός κίνδυνος, είναι η πείνα, η φτώχεια στον κόσμο. Κοιτώντα λοιπόν τη Μεσόγειο ή αλλού στον κόσμο, αλλά στη Μεσόγειο γιατί ευθύνη πιο κοντά μας, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους που δεν ξέρουν να κολυμπάνε, που μπαίνουν πάνω σε σκάφη, σχεδίες, οτιδήποτε, για να φτάσουν στις ακτές της Ιταλίας, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι συχνά σοκάρομαι που ακούω υπεύθυνους, πολιτικούς, σε υψηλές θέσεις που λένε ότι εμείς όταν θα είμαστε στην κυβέρνηση δεν θα υπάρχει πια μετανάστευση. Πολύ δύσκολο όμως είναι αυτό, γιατί εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να εμποδίσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, να προσπαθήσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο. Είναι τα δημόσια αγαθά αυτά που λείπουν από τους πληθυσμούς αυτούς. Και ποια είναι αυτά? Είναι πόσιμο νερό, είναι τρόφιμα, είναι το δικαίωμα, η πρόσβαση στις θεραπείες, στα φάρμακα, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Αν θέλουμε από εκεί και πέρα να αναπτύξουμε προγράμματα, οικονομικά προγράμματα, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτά τα αγαθά, τα παγκόσμια αγαθά όπως τα λέω εγώ, τότε δεν θα πετύχει τίποτα. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια βλέπουμε ότι έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που κερδίζουν κάτω από 1,25 δολάρια. Και αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παγκόσμια αγαθά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσω αυτού του μηχανήματος ενημερώνονται όλο και περισσότερο για τον πλούτο που υπάρχει λίγα χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκονται οι ίδιοι. Συνεπώς η κατάσταση γίνεται έτσι εκρηκτική και για τη μετανάστευση αλλά και για τους εξτρεμισμούς οι οποίοι τροφοδοτούνται από τέτοιου είδους απελπισία που πλήττει τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι οι δωρητές χώρες, οι χώρες του ΟΣΑ χοντρικά, είναι χώρες που πλήττονται από οικονομική κρίση και σημαντική δημοσιονομική κρίση. Η δικιά μου, για παράδειγμα, είναι ένα παράδειγμα. Ο προπολογισμό δυσκολεύεται όλο και πιο πολύ. Οι ακραίε θέσει ανεβαίνουν. Πολλοί άνθρωποι εκφράζουν δυσαρέσκεια. Και όταν του ζητάμε να δώσουν περισσότερα για αυτού που βρίσκονται 4-5 χιλιόμετρα πέρα από αυτού, λένε Μα και εμεί υποφέρουμε. Οπότε τι θέλετε. Συνεπώ, η δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη μειώνεται. Πέρα από κάποιε βόρειε χώρε, τη Βόρεια Ευρώπη δηλαδή, τον οποίο τη βοήθεια χαιρετίζω πραγματικά η αναπτυξιακή βοήθεια προς τον τρίτο κόσμο μειώνεται συνεχώς. Συνεπώς καταλήγουμε. Απ' τη μια οι ανάγκες να αυξάνονται ραγδαία για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να βρεθεί πόσο βοήθεια κτλ. Και απ' την άλλη μεριά τα έσοδα μειώνονται. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αντιδράσουμε. Και πώς με καινοτόμα χρηματοδότηση προς την ανάπτυξη. Υπάρχουν πέντε οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες εποφελούνται από την παγκοσμιοποίηση. Είναι ο μαζικός τουρισμός με τις αεροπορικές μεταφορές, είναι οι οικονομικές συναλλαγές με τους μαθηματικούς αλγόριθμους. Σήμερα έχουμε ε, χιλιάδες ανά δέκατο δευτερολέπτου τέτοιες συναλλαγές. Έχουμε το διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια στα χρηματιστήρια Αυτά τα αυτές οι εταιρείε ανέβηκαν περισσότερο, που πληρώνουν βέβαια χαμηλούς φόρους σε φορολογικούς παραδείσους. Τέταρτον είναι η κινητή τηλεφωνία και πέμπτον είναι η εξορρυκτική πόρη. Για να τελειώσω πρόεδρε και για να αρχίσει έτσι η συζήτηση, δύο παραδείγματα θα σας δώσω. Το 2006 με τον πρόεδρο Σιράκ, ο πρόεδρος Λούλα, ο Λάγκος της Χιλής και ο κύριο Μπανκιμούν, που ήταν υπουργό εξωτερικών της Νότιας Κορέας τότε, φέραμε μια ιδέα. Ένα δολάριο ή ένα ευρώ ανά εισιτήριο αεροπορικό. Έγινε συζήτηση λοιπόν στο, στη Βουλή, στη Γαλλία και πολλοί άνθρωποι είπαν ότι για άλλη μια φορά η Γαλλία θέλει να αλλάξει τον κόσμο και θέλει να δώσει μαθήματα στους πάντες. Εμείς με άλλες χώρες πετύχαμε, 13 χώρες συνολικά, όντως ένα ευρώ ή ένα δολάριο να παίρνουμε από κάθε αεροπορικό εισιτήριο. Ένας νόμος ήταν αυτός, ήταν σαν μια υποχρεωτική εισφορά. 2 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια δολάρια μαζέψαμε σε 7 χρόνια. Και αποφασίσαμε να αγωνιστούμε με τον έκτο στόχο που ήταν ακριβώς να αντιμετωπιστεί η θυματίωση, η ελαιονοσία κλπ είναι μια μικρή ιδέα. 8 στους 10 σήμερα θεραπεύονται. 8 στα 10 θεραπεύονται χάρη σε αυτή τη βοήθεια που μπορεί να είναι μικροσκοπική σε σχέση με το σύνολο της αλληλεγγύης που χρειάζεται να επιδείξουμε. 350 εκατομμύρια ε, θεραπείες χρηματοδοτήθηκαν για την ελαιονοσία και 2,5 εκατομμύρια παιδιά για τη φημετίωση. Είναι λίγο, πολύ λίγο. Αλλά δείξαμε στον κόσμο ότι μια τόσο μικρή ένδειξη αλληλεγγύης μπορεί να κάνει τα πράγματα να αλλάξουν. Γιατί δεν είναι γνωστά όλα αυτά. Γιατί δεν έχουμε μπλουζάκια, δεν έχουμε κασκέτες που να τα λένε όλα αυτά, αλλά χρηματοδοτούμε τη UNICEF, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και μεγάλες ε, τέτοιες οργανώσεις. Δεύτερο παράδειγμα στην Αντίσα Μπέμπα, πολύ σύντομα. Θα έχουμε το Unit Life. Πείσαμε έξι Αφρικανούς ηγέτες να δώσουν δέκα σαντίμ για κάθε βαρέλι δολάριο ή αντίστοιχα για χρυσό ή για ουράνιο. Οι πόροι αυτοί λοιπόν, οι πρώτες ύλε που βρίσκονται σε αυτές τις τυχερές χώρες που έχουν τόσο πλούσιο υπέδαφος μπορεί να βοηθήσει στην αλληλεγγύη αυτή για την καταπολέμηση τη, του λοιμού. Πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο υποφέρουν με φοβερές συνέπειες στον εγκέφαλό τους. Γι' αυτό και τόσο δύσκολα προχωράει στην ανάπτυξη μια τέτοια ήπειρος όπως είναι η Αφρικανική, η Ινδία. Αυτά ήθελα να πω εισαγωγικά. Αρκεί δηλαδή να θέλει κανείς, να θέλουν οι επικεφαλής κατών και κυβερνήσεων. Χρειάζεται αυτή η βούληση τότε μπορούν να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν και να ζητήσουν από την κοινή γνώμη να πιέσει. Και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ βέβαια για άλλη μια φορά που με προσκαλέσατε. Υπάρχουν και άλλα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μικροσκοπικός φόρος 0,01 για κάθε παράγωγο, χρηματοοικονομικό παράγωγο. Κανεί δεν θα το καταλάβει. Κι όμως θα άλλαζε έτσι η εξέλιξη στον κόσμο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Για να αρχίσουμε τη συζήτηση, κυρία Λιωμαρή πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα, Πρόεδρε, με τη σειρά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ξαναβλέπω τον Φιλίπ του Πλασί, που γνωρίζω πόσο αφοσιωμένος είναι σε όλα αυτά τα θέματα εδώ και χρόνια. Και με αυτή τη δράση απέδειξε ότι όταν θέλουμε κάτι μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο μάθημα που πρέπει να συγκρατήσουμε σε έναν κόσμο που πολύ συχνά υπάρχουν καλά λόγια και δεν δίνεται συνέχεια όσον αφορά την υλοποίησή τους, κυρίως όσον αφορά την οικονομική υλοποίηση των αποφάσεων, νομίζω ότι σήμερα έχουμε ένα καλό παράδειγμα τι θα έπρεπε να κάνουμε. Θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είναι προφανές ότι το AIDS είναι ένα πρόβλημα σημαντικό για την Αφρική, όμως η UNITAID ασχολείται εξίσου και με άλλες υπήρους η ιδέα είναι να επικεντρωθείτε επί της Αφρικανικής Υπήρου ή μήπω υπάρχει κάποιο άνοιγμα, διότι αυτό που με εντυπωσιάζει, κυρίως όσον αφορά το πρόβλημα της μετανάστευσης σήμερα, είναι ότι η μετανάστευση εξίσου συνδέεται στενά με την αστάθεια κάποιων χωρών και ξεφεύγουν από το θάνατο κάποιοι οι άνθρωποι αυτοί. Και εγκρίνω αυτά που είπατε προηγουμένως, δηλαδή όταν κάποιοι δεν έχουν παρά μόνο την εναλλακτική να πεθάνουν επί τόπου ή να ρισκάρουν τη ζωή τους για να πάνε σε χώρες που τους φαίνονται πιο ασφαλείς και όπου θα εξασφαλίζουν τα ελάχιστα προς επιβίωση και να μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους, είναι προφανές ότι θα εξακολουθούν να το προσπαθούν. Αλλά έχουμε την έκρηξη της ε, ανασφάλειας, των συγκρούσεων, των εντάσσεων στην Αφρική και των κινδύνων, στην Εγγύης Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, είναι προφανές ότι αυτό το φαινόμενο της μεταναστεύσεως θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Και δεν μπορούμε να προσπαθούμε να συγκρατήσουμε στην άφηξη τα μετασταυτικά κύματα, αλλά καλύτερα θα μπορούσαμε να κινηθούμε σε διπλωματικό επίπεδο, να κινηθούμε στις ρίζες της μετανάστευσης εάν κινηθούμε στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο βοηθώντας ε, να έχουν ανάπτυξη οι πληθυσμοί αυτοί και να βοηθήσουμε την υγεία τους. Η δράση της UNITED πώς εντάσσεται σε ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να είναι αναγκαία ευρύτερο και βέβαια εξυπακούεται όλες οι εμπλεκόμενες χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν. Η Ευρώπη, αλλά όχι μόνο η Ευρώπη, διότι κάθε χώρα που φαίνεται ότι είναι πιο πλούσια, πιο ασφαλής από ό,τι γειτονική, αυτόματα θα προσελκύσει μια μετανάστευση που μπορεί να την αποσταθεροποιήσει και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πλάνκοβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην περίοδο που ήμουνα σε μια θέση στο Παρίσι που ήσασταν Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας και θυμάμαι τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Σιράκ που πραγματικά είχε καταβάλει προσπάθειες να επεξεργαστεί την έννοια αυτή της αλληλεγγύη για να βοηθήσει τους πλέον στερημένου και τους έχοντες ανάγκη. Και είμαι ικανοποιημένο που άκουσα την ανάλυση σας, που τόσα πολλά χρήματα συνελέχθησαν βάσει της ε, πρωτοβουλίας με ένα ευρώ ή ένα δολάριο κατά εισιτήριο αεροπορικό. Μεγάλη πρωτοβουλία που ήδη χρονολογείται το έτη. Λοιπόν, αυτή τη συνεργασία με τους μεγάλους χρηματοδοτικούς φορείς, ε, ποιος ο ρόλος ή η συνεισφορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να, πώς μπορεί να είναι πιο ορατή, πιο συγκεκριμένη η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ, ο κύριος Πεγιούν έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Γενικέ Γραμματεύ αναπληρωτή Γενική Γραμματεύ, θα ήθελα να πω ότι το κείμενό σα είναι αξιοσημείωτο, πολύ ισχυρό, αλλά κάπου πάσχει όσον αφορά τον φόρο για τις μοτοστατικές συναλλαγές. Χρονολογείται αυτή η προσπάθεια από παλιά, εδώ και 20 χρόνια. Τη λιδόρισαν εδώ και 20 χρόνια. Σε αυτό το κοινοβούλιο, στην προηγούμενη θητεία, είχαμε ετοιμάσει ένα κείμενο που ετοίμασαν κάποιοι βουλευτές και ήταν πολύ δύσκολο να εγκριθεί πάντα έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε μείνει 20 χρόνια πίσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δυσκολίε και βλέπω διαπραγματεύσει όσον αφορά το κλίμα θα είναι ένα από τα αίτια όσον αφορά την Αφρική για τα προβλήματα και βλέπουμε με πόση δυσκολία και με πόσο αργό ρυθμό ο εκτελεστικός κλάδος κινείται για να ανταποκριθεί στο ύψο των περιστάσεων. Υπάρχει ένα είδο πολιτική μοιοπίας που κοστίζει πολύ ακριβά στις οικογένειε μα και στι χώρε μα. Έχω δύο ερωτήσεις ε, όσον αφορά αυτά που μας λέτε και τα οποία χαιρετίζω ε, εκ βαθέων. Είναι μια προπτική και θα πρέπει να ενωθούμε στην προπτική. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η θέση. Είσαστε γιατρός εσείς και ήσασταν αξιοσημείωτος στο έργο που κάνατε όσον αφορά το AIDS και την ονοσία. Ποια είναι η θέση της παιδείας, της εκπαιδεύσεως, θα αναφέρετε επανειλημμένα στο κείμενό σας. Γίνονται πολλές συζητήσεις στη Γαλλία όσον αφορά τη σχετική μας συνεισφορά, όσον αφορά την παιδεία και την υγεία. Και εγώ ασχολήθηκα με το θέμα. Πώς βλέπετε εσείς αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τις αφρικανικές χώρες για τη συνεργασία στον τομέα τη παιδείας. Δεύτερον, στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την κατανομή των εσόδων των φορολογικών. Μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα για να εφαρμοστεί αυτό το θέμα. Δεν συμμετέχουν οι χώρε. Ε, δημιουργούνται στευλώσει του ανταγωνισμού και αυτό είναι πάρα πολύ ενσυχητικό. Ταυτόχρονα όμω ε, κάποιοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, και ο Πρωθυπουργό τη Ισπανία και τη Γαλλία θέλουν αυτή η φόρη τα έσοδα να διατίθενται και κάποιε οτεραιότητε. Ε, Ποιε προσπάθειε καταβάλλονται, είναι πολλέ, κυρίω ποιο ποσοστό, για ποιο ποσοστά μιλάμε. Ένα ποσοστό τον φόρο να διατίθεται, αλλά ποιο. Διότι είναι ακόμα πολύ μικρά τα ποσά, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα διάφορα δικηβεύματα. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε από αυτού και σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε. Ο κ. Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Θέλω και εγώ να σα καλωσορίσω εδώ, αγαπητέ κύριε, και να ευχαριστήσω πρωτίστω για όλο τον κόπο που κάνετε για άμβλυνση των προβλημάτων με τα οποία ασχολείστε. Είπατε ε, πάρα πολύ σωστά ότι μερικοί παράγοντες συμβάλλουν στο να έχουμε τεράστια μετανάστευση, η έλλειψη νερού, είπατε, τροφίμων, πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση. Πάρα πολύ σωστά. Ε, θέλω να επισημάνω ότι λείπει κάτι από αυτή την προσέγγιση που είναι ίσως ο θεμελιός των προβλημάτων στα οποία αναφέρεστε και που είναι οι πόλεμοι και οι πόλεμοι δημιουργούνται από κάποιους. Ε, μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα πώς δεν το θίξατε και δεύτερο, εάν βλέπετε ότι η δημιουργία πολέμων, κυρίως στις περιοχές από όπου προέρχεται η μετανάστευση, είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και το αφήνουμε απλώς έξω. Θεωρώ δηλαδή ότι η ασφάλεια Βεβαίω το νερό, τα τρόφιμα, η πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, χωρί καμιά συζήτηση, τεράστια σημασία. Αλλά πάνω απ' όλα δεν είναι η ασφάλεια. Μπορεί να είμαι σε μια περιοχή και να ζω πάρα πολύ φτωχά και να νιώθω και σχετικά ευτυχισμένο εάν έχω ασφάλεια. Και θέλω έτσι να αναλύσετε λίγο αυτή την απουσία προσέγγιση αυτή τη ψυχή του προβλήματο. Ευχαριστώ. Señor Epitideos. Κύριε Πιτίδιο. Κύριε Πρόεδρε, ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον 21ο αιώνα που ζούμε υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες κάθε άλλο και κολακευτικές είναι για τον δυτικό πολιτισμό και αποτελούν την αιτία της ε, του, σημερινού κύματος μεταναστεύσεως. Όμως, η φιλοσοφία ότι επειδή υπάρχει δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι, έχουν προβλήματα στις χώρες τους, να βλέπουν ότι οι γειτονικέ χώρε είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να πάνε σε αυτέ και να μείνουν εκεί δεν διαφέρει καθόλου από την φιλοσοφία που είχαν οι πειρατέ πριν μερικού αιώνε. Και αυτοί έβλεπαν κάποια πλοία πλουσίων χωρών ή κάποιε χώρε που ήταν πλούσιε και εισέβαλαν εκεί. Μια τέτοια φιλοσοφία δεν πρέπει να επικρατεί η σημερινή εποχή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τι ρίζε του προβλήματο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε οικονομικά τις χώρες αυτές. Να έχουμε δημοκρατικές κυβερνήσεις εκεί. Να μην επιτρέπουμε την εκμετάλλευση των λαών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την εκμετάλλευση των οικονομικών πόρων των περιοχών αυτών προς όφελος των χωρών εκείνων. Και όταν στέλνουμε κάποια οικονομική βοήθεια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθεια αυτή δεν θα πάει σε διασταρμένες κυβερνήσεις αλλά στο λαό κάθε χώρα που έχει ανάγκη. Θα ήθελα λοιπόν να μας αναπτύξετε, πολύ περιληπτικά βεβαίως, ε, ποια είναι η προσπάθεια συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΗΕ προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Eh, κύριε ευχαριστώ πολύ κύριε Δεπλασί που ήρθατε. Θέλω να σας δείσω περισσότερο περισσότερες πληροφορίες για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εμείς και η χώρα μου η Ισπανία συμφώνησαν. Αλλά θέλω να ξέρω ποιες άλλες χώρες από τη διεθνή κοινότητα στηρίζουν αυτή την πρόταση. Έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ. Και μέσα σε αυτές τις καινοτόμες ιδέες χρηματοδότησης που είναι πολύ σημαντικές τώρα που βρισκόμαστε σε κρίση πολλές χώρες, Πώς βλέπετε τις προοπτικές που υπάρχουν για την ατζέντα μετά το 2015 που θα καθοριστεί στη Νέα Υόρκη το φθινόπωρο. Εσείς πώς βλέπετε τη διαδικασία που ακολουθούμε για να καθοριστεί αυτή ακριβώς η ημερήσια διάταξη μετά το 2015. Ο κύριος Παντσέρη τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Υπογραμμίζω και εγώ τη σημασία που έχει η δραστηριότητά σας και ο ρόλος που παίζετε, διότι η λήψη ενός συνολικού πλαισίου και δυνατότητας παρεμβάσεως μέσω ανθρωπιστικής συνεργασίας και βοηθείας ε, δεν θα λύναμε τα προβλήματα. Είναι σημαντικό. Έχω δύο ερωτήσεις. Πιστεύω ότι αναφυσβήτητα γνωρίζετε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που περιγράψατε αν δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα αίτια, θα έχουμε τελικά ένα πίθμενο πηγάδι στα χέρια μας. Έχω συχνά την εντύπωση ότι το, η δεξιά χείρ του ΟΗΕ δεν γνωρίζει την πράτη αριστερά. Είναι σημαντική πτυχή της δραστηριότητα που εφαρμόζει ο ανθρωπιστικός ΟΗΕ και όμως δεν επηρεάζει πολύ τον πολιτικό ΟΗΕ. Είναι θεμελιώδες αυτό διότι είναι τελικά σαν το σκύλο που δαγκώνει την ουρά του. Ένας ουροβόρος. Λοιπόν, δεύτερο στοιχείο. Ποια είναι η πολιτική συνεργασία. Και αν αναφέρουμε την Αφρική γνωρίζετε άριστα ότι είναι, ε, είναι, ε, έχει μεγάλα προβλήματα η Αφρική. Ε, και έχουμε και προβλήματα να λύσουμε τις, τα προβλήματα συνεργασίας. και έχουμε και ανταγωνισμό με χώρε άλλε, όπω είναι η Κίνα που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Κίνα στην Αφρική. Πώ εντάσσεται η δραστηριότητα της συνεργασίας και της βοηθείας του ΟΗΕ διότι το κομβικό σημείο μεταξύ δημοκρατίας ε, και ε, βοηθείας είναι πολύ σημαντικό κόμβο. Κινδυνεύουμε να δίνουμε χρήματα εκεί που υπάρχουν οι διάφορα δεσποτικά καθεστώτα που και έτσι δεν παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει αυτός ο προβληματισμός ούτως ώστε η ίδια η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιο τρόπο να συμπληρώνει και να επικουρεί τις δραστηριότητες που έχετε υπόψη κυρίως όσον αφορά την Ήπειρο την Αφρικανική. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας για αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζιουβέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε αναπληρωτή Γενική Γραμματεύ. Σας ευχαριστώ πρώτα για την παρουσίαση του θέματος που δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε τώρα μια διπλή επιταγή, αφενός μια ηθική επιταγή προφανή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ο κόσμος να συνεχίζει να πλουταίνει από τη μια μεριά και να φτωχαίνει από την άλλη. Μια ηθική επιταγή λοιπόν. Κυρίως λοιπόν αυτό. Αλλά είναι και το δικό μας το συμφέρον οι μεταναστευτικές πιέσεις, τις οποίες αναφέρθηκαν ήδη ορισμένοι, είναι πραγματικές και είναι και πολιτικό θέμα. Η πρόθεση λοιπόν εργαλείων, όπως αυτή η καινοτομία για την ανάπτυξη, μπορεί να, να ανταποκρίνεται και σε μια ηθική επιταγή, αλλά και στο ίδιο συμφέρον των ευρωπαϊκών χωρών. Μια απλή ερώτηση, ίσως και λίγο απλοϊκή. Γνωρίζετε κύριε Γενική Γραμματεύ ποιες είναι οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε ποιες είναι και ποιες μπορούν να είναι οι αρμοδιότητές του που είναι λίγες όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απομονωμένο χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς τις χώρες μέλη ιδίω είναι αδύνατον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει μόνο του μια πολιτική. Ωστόσο, αν είχατε μία ευχή να μπορείτε να την εκφράσετε εδώ, που να αφορά μονάχα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού θα μπορούσε να σας βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο καθήκον σας να σας διευκολύνει για την εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης σε ευρεία βάση, για να μπορέσετε να κάνετε όσο γίνεται περισσότερα. Ευχαριστώ. Η τελευταία ερώτηση είναι δική μου. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σε τι επίπεδο πόρων βρισκόμαστε για να πετύχει ένα σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Και εσείς πώς θα αντιλαμβάνεστε, πώς νομίζετε ότι πρέπει να δράσουμε ώστε να έχουμε ένα πραγματικό αντίκτυπο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ερωτήσεις σας. Γιατί όλοι θέσατε πολύ εύστοχα ζητήματα. Υπάρχουν τρεις παγκοσμιοποίησεις θα έλεγα της οικονομίας που έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ εξαιτία του διαδικτύου και μας μένει η τρίτη που λείπει ακόμα και είναι η παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης. Η πρώτη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έγινε από τους επιχειρηματίες. Οι οποίοι τι θέλουν την παγκοσμιοποίηση. Δεν περνάει από το μυαλό κάποιο επιχειρηματία ότι θα πουλάει μόνο στην Ισπανία, μόνο στη Γαλλία. Όχι. Θέλει να έχει όλο τον κόσμο στη διάθεσή του. Η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας επίσης έγινε από τους επιχειρηματίες. Όμως εξαρτάται και από τους πολιτικούς και από εμά. Οι πολιτικοί Δυστυχώ όμω ενδιαφέρονται για το τοπικό επίπεδο και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτού. Οι πολιτικοί κοιτούν μόνο τι εκλογέ που θα γίνουν μετά από 2-3 χρόνια. Εννοείται ότι δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές αν μιλήσουμε στον κόσμο μας για τα μεγάλα θέματα για τα οποία μιλάμε εμείς εδώ σήμερα. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να αποφασίσουμε ότι η πολιτική σημαίνει το τι θα γίνει τα επόμενα 15-20 χρόνια. Και αυτό είναι το σημερινό ζήτημα. Η παγκοσμιοποίηση τη αλληλεγγύη. Σήμερα το πρωί από το Reuters, από το AFP, είχαμε κάποια νέα που λένε ότι 16% παραπάνω στον κόσμο των εκατομμυριούχων έχουμε. Υπάρχει δηλαδή σήμερα ένα σύστημα με ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους στοχούς που δεν καταφέρνουμε να κλείσουμε. Η κυρία Λιωμαρή έθεσε ένα ερώτημα σημαντικό. Λέει για τη δουλειά που γίνεται στην Αφρική, αν υπάρχει κάποια μονάδα που δουλεύει για την Αφρική ειδικά. Όχι, για τις πιο φτωχές χώρες που υποφέρουν από το AIDS, την ελονοσία κλπ. και θυματίωση. Όταν μιλάμε για παιδιά με AIDS, το 98% αυτών των παιδιών είναι στην Αφρική. Το 99% των γυναικών που βρίσκονται, στην, που έχουν μάλλον AIDS, είναι στην Αφρική. 80% της ελονοσίας είναι στην Αφρική. Γι' αυτό είμαστε κύρια στην Αφρική. Γιατί αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτές τις τρεις ασθένειες. Η κυρία Λιωμαρή επίσης ρώτησε κάτι άλλο σημαντικό. Όπως και κάποιος άλλος ευρωβουλευτής. Ρωτήσατε για τους πολέμους. Ο κύριος Χατζηγεωργίου για παράδειγμα και η κυρία Λιωμαρή ρώτησαν για τον πόλεμο. Ε, λέτε, μιλάτε για την πείνα, για το πόσιμο είδωρ, για την υγεία, την εκπαίδευση. Λέτε ότι γι' αυτό φεύγει ο κόσμος. Μα όχι, φεύγει εξαιτία του πολέμου, λέτε. Εδώ θέλω να σας μεταφέρω κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος. Ότι η άκρα ένδια, φτώχεια δηλαδή, πάντα έχει κάποια συνέπεια και είναι πάντα ίδια. Περισσότερη βία, περισσότερες σειράξεις, περισσότεροι πόλεμοι. Όταν κάποιος είναι πάρα πολύ φτωχός, όταν ένας λαός υποφέρει από φτώχεια, αμέσως υπάρχουν συγκρούσεις. Συνεπώς, υπάρχει άμεση σχέση, αναλογική και προφανής ανάμεσα στην άκρα φτώχεια και τη βία. Λέμε συχνά και υπάρχουν πολλοί θαραλέοι που λένε ότι άμα φροντίσουμε για το AIDS, την αλλονοσία, τη τα κτλ, θα είμαστε 15 δισεκατομμύρια πάνω σε αυτή τη γη. Πώς θα γίνει. Ναι, όταν μια γυναίκα, ένα ζευγάρι σε μια πολύ φτωχή χώρα κάνουν παιδιά, η παιδική θνησιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνουν 8 παιδιά για να τους μείνουν 4 που θα μεγαλώσουν αν ο πλούτος της χώρας αυξηθεί, τότε θα κάνουν και λιγότερα παιδιά. Αυτό το είδαμε στην Αλγερία, στην Τινησία, στο Μαρόκο σήμερα. Αν αυξήσετε την οικονομική ανάπτυξη σε μια χώρα, θα μειωθεί η άκρα φτώχεια. Και γι' αυτό αυτά που είπε ο κύριος Πηγιό ισχύουν. Είναι η εκπαίδευση, ναι. Από τη στιγμή που θα έχουμε σχολεία, από τη στιγμή που θα δώσουμε εκπαιδευτικές αξίες στα παιδιά, τότε αμέσως θα αλλάξει η διακυβέρνηση, ε, θα βλέπουμε αλλιώ τον άλλον, θα σεβόμαστε τον άλλο περισσότερο. Είναι το θέμα της νοοτροπίας, που δεν είναι ίδιες βέβαια παντού ευτυχώς, αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στη διαφορά τους αυτές οι νοοτροπίες όλες να σέβονται τον άλλον. Έχετε δίκιο και η κυρία Λιωμαρή επίσης και ο κύριος Χατζηγεωργίου για το ότι οι πόλεμοι κάνουν τον κόσμο να φεύγει από τις χώρες του, αλλά πίσω από τους πολέμους υπάρχει άκρα φτώχεια. Κύριε Πλάκοβιτς, η εταιρική σχέση Ηνωμένα Έθνη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η Ευρώπη κάνει πολλά. Κάνει πολλά στις πιο φτωχές χώρες, χωρίς να το γνωστοποιεί όμως. Και είναι κρίμα. θα λέγω ότι δεν προωθείται επαρκώς η πολιτική αυτή από τα ίδια τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ίσως γιατί δεν υπάρχει ένας κύριος Ευρώπη που να εκλέγεται, δεν ξέρω γιατί, πιστεύω ότι είναι κρίμα, αλλά έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήπειρος που κάνει τα περισσότερα με την Αμερική για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν προβάλλεται. Η εταιρική σχέση είναι προφανές ότι βοηθάει. Θα ήθελα να έχουμε εταιρική σχέση μεταξύ της Unit Unit Life και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Και γιατί, θα σας πω γιατί. Κάναμε κάτι που είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου που έγινε. Και αυτό είναι ότι σήμερα 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν συμμετέχουν στην ιατρική πρόοδο. Υπάρχουν ε, άνθρωποι που πεθαίνουν, του δείχνουμε το φάρμακο, του λέμε κοίτα, να υπάρχει το φάρμακο αλλά δεν είναι για σένα. Γιατί, Γιατί τα φάρμακα αυτά είναι στι πιο πλούσιε χώρε και για 15-20 χρόνια προστατεύονται από διπλώματα ευρωσιτεχνίας. Οι υπόλοιποι, τα 2 δισεκατομμύρια πεθαίνουν γιατί δεν έχουν στη διάθεσή του αυτό το φάρμακο. Για το AIDS λοιπόν έχουμε ένα σύστημα που είναι μια κοινότητα διπλωμάτων ευρεσιτεχνία που επιτρέπει στου πιο φτωχούς για πρώτη φορά στην ιστορία να έχουν στη διάθεσή του τα ίδια φάρμακα με τους πιο πλούσιους αλλά 80% πιο φθηνά. Medicine Main Pool λέγεται. Ψάξτε το στο Google, ψάξτε το και σε άλλες ιστοσελίδε. Είναι η πρώτη φορά που με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτρέψουμε στου πιο φτωχού να έχουν στη διάθεσή τους τα ίδια φάρμακα. Για το θέμα αυτό, κύριε Πλένκοβιτ, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγο. Για αυτά τα θέματα μπορεί να κάνει κάτι. Ένα φάρμακο, όπως αυτό το, σακάκι. Αυτό το σακάκι μπορώ να το αγοράσω σε αυτή τη τιμή. Αν δεν μπορώ να το αγοράσω σε αυτή τη τιμή, να το αγοράσω πιο φθηνά. Δεν είναι σοβαρό, αν δεν μπορώ. Το φάρμακο όμως είναι. Αν υπάρχει το φάρμακο και εγώ θα πεθάνω επειδή δεν μπορώ να το έχω, ε, είναι μεγάλη αμαρτία και είναι ένα θέμα της ανθρωπότητας ολόκληρης. Αυτό το σύστημα πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλο τον κόσμο. Οι τιμές για την υπατήτηδα γάμα. 85.000 για να σωθεί ένας άνθρωπος ενώ κοστίζει 25 δολάρια. Είναι φοβερό. Είναι ένα θέμα που η διεθνής κοινότητα θα κληθεί να αντιμετωπίσει μέσα στα επόμενα χρόνια. Φυσικά και υπάρχει το χρηματιστήριο. Φυσικά και υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Εννοείται. Αλλά είμαστε πολιτικοί. Πρέπει να είμαστε πάνω από όλα αυτά, υπεράνω. Ε, με ρωτήσατε και ο κύριος Μιχαμούν και άλλοι για τον φόρο συναλλαγματικών ε, συναλλαγών, ε, συναλλαγών. Δεν μπορούν να αποφασίσουν όλες οι γενιές ότι 0,01% αλλάζει τον κόσμο. Αν πάρουμε 0,1% και 0,01% από χρηματοπιστωτικό παράγωγο σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε 400 δισεκατομμύρια στον κόσμο. Και έτσι απαντάω και στην ερώτηση του Προέδρου που ρωτάει πόσα χρειάζονται για να αποφύγουμε αυτά τα δράματα, αυτές τις τραγωδίες. Το ερώτημα δεν είναι αν θα ισχύσει αυτός ο φόρος. Θα δείτε. Πριν από 20 χρόνια ήμασταν πολύ λίγοι που θέλαμε αυτόν τον φόρο χρηματοπιστατικών συναλλαγών είχαν πει δεν γίνεται, εσύ είσαι γιατρός, δεν ξέρει τίποτα από την οικονομία, δεν είναι εφικτό. Σήμερα ήδη μας λένε είναι εφικτό. Το πρόβλημα είναι ότι είναι εφικτό για τους εθνικού προπολογισμού και διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες κυβερνήσει, τα ίδια Υπουργεία Οικονομικών βρίσκουν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά αν κρατήσουν τα χρήματα. Η συζήτηση γίνεται σε διάφορες χώρες. Στη Γαλλία η κυβέρνηση δέχτηκε να δώσει 30% του προϊόντος αυτού, του φόρου δηλαδή αυτού, κάτι που είναι ιστορική σημασία. Ο Υπουργό Οικονομικών θεώρησε ότι είναι πολύ και μείωσε άλλα ποσά τα οποία δίνονται στην ανάπτυξη. Εν πάση περιπτώσει πηγαίνει το 30% του φόρου αυτού στην ανάπτυξη. 11 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ισπανία και η Γαλλία το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να υπάρχει ένας τέτοιος φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών. Το θέμα είναι να δούμε τώρα πώς θα πιέσουμε ώστε οι Υπουργοί Οικονομικών να δεχτούν να δώσουν τουλάχιστον 30 με 50% του φόρου αυτού στην ανάπτυξη. Πολιτική μοιοπία υπάρχει. Ναι, Συμφωνώ με τη διατύπωση αυτή. Ο κύριος Μίγιαμαν ρώτησε ποιες είναι οι άλλες χώρες. Στην Ταϊλάνδη σήμερα έχετε μεγάλες συζητήσεις για το φόρο αυτό χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και στη Βραζιλία, κύριε Μαρουσέφ το έκανε, που απευθύνεται όμως μόνο στην υγεία. Και για την υγεία στη Βραζιλία Οπότε, ακόμα γίνεται η συζήτηση για τον φόρο αυτό και την ανάπτυξη. Βεβαίως, το 2017 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά κύριε Μηγιαμένη. Το λέω στο Κοινοβούλιο, το 2017 είναι σημαντική χρονιά γιατί είναι η χρονιά όπου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα παρουσιάσουμε το Sustainable Development Goals, τους στόχους δηλαδή βιώσιμης ανάπτυξης είναι το τέλος των στόχων της χιλιετίας και η αρχή των στόχων της βιώσιμης χιλιετίας. Και εδώ έχετε βέβαια απόλυτα δίκαιο που επιμένετε. Αν θέλουμε να είμαστε σε αυτό το ραντεβού, πρέπει να είμαστε και στο ραντεβού για τις καινοτόμες μεθόδους χρηματοδότησης. Και έρχομαι τώρα στη χρηματοδότηση, στην, στην εκπαίδευση. Ποιος είναι ο ρόλος της παιδείας, της εκπαίδευσης. Ρωτήσατε κάποια πράγματα και όντω είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να έχουμε καινοτόμα χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και γιατί είναι τόσο εύκολο να έχουμε καινοτόμα χρηματοδότηση για την υγεία. Όταν λέμε ότι 8 στα 10 παιδιά τα θεραπεύουμε από το AIDS, είναι 8 στα 10, έτσι, με νούμερα, μπορούμε να το ξέρουμε. Στην εκπαίδευση πώς να το εκφράσουμε αυτό ποσοτικά. Αυτό είναι η δυσκολία. Έπειτα για τον κύριο Επιτίδιο καλή διακυβέρνηση στις υπονάπτυξη χώρας. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό μιλάω για την εκπαίδευση. Αν εκπαιδευτούν τα παιδιά θα υπάρχει και καλύτερη διακυβέρνηση. Κύριε Παντζέρη, κάνει το δεξί χέρι του ΟΗΕ κάτι και το αριστερό κάνει κάτι άλλο. Μα ποιος είναι ο ΙΕ. Ο ΙΕ δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΙΕ είναι το αποτέλεσμα των όσων κάνουν όλε οι χώρε του κόσμου. Και κυρίω. Εκείνε που βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Και αυτό πρέπει να πούμε στα εκτελεστικά μας όργανα. Μην κάνετε με το δεξί κάτι διαφορετικό με αυτό που κάνετε με την αριστερά. Είναι σωστό. Και το δεξί και το αριστερό χέρι πρέπει να κάνουν το ίδιο, προ την ίδια κατεύθυνση. Έχετε δίκιο για το ότι οι Κινέζοι δίνουν χρήματα διμερώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το κάνει. Σήμερα πρέπει να επικοινωνούμε περισσότερο για τα χρήματα που δίνουμε στις πιο φτωχές χώρες, να γίνεται γνωστό. Και θα τελειώσω με τους δύο τελευταίους που πήραν τον λόγο. Πρόεδρε, ρωτάτε πόσα η αναπτυξιακή βοήθεια έχει περάσει από 100 136 δολάρια το χρόνο. Για τα ζητήματα υγείας και εκπαίδευσης 50 δισεκατομμύρια το χρόνο χρειάζονται ακόμα, που δεν είναι τίποτα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα που χρειάζεται τη βοήθεια. Κλιματικές αλλαγές. 100 δισεκατομμύρια το χρόνο, λέει Κοπεχάγη. Δεν έχουμε φτάσει στα 10 ακόμα. Και λίγες μέρε μας χωρίζουν από το Παρίσι. Και θα τελειώσω με αυτό που είπε ο κύριο Ζουβά. Ποια είναι η ευχή, η επιθυμία του σώματος στο οποίο ανήκω. Η επιθυμία που μπορώ να εκφράσω είναι η ευρωπαϊκοί λαοί που εκπροσωπείτε, εσείς οι ευρωβουλευτές, να κάνετε έκκληση προς όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου για να πείτε ότι τώρα που είμαστε λίγες μέρες πριν από το COP21, τη Διεθνή Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα, λίγες μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΙΕ, όπου θα παρουσιάσουμε τους στόχους της ε, αηφόρου ανάπτυξη, να πείτε ότι η μόνη λύση για να αποφεύγουμε παγκόσμιο πόλεμο τον 21ο αιώνα είναι να βρούμε τέτοιες μικρές δράσεις αλληλεγγύης για ε, να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Τέτοιε κοινοτόμε λύσεις χρειάζονται και είναι το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε εν ειρήνη τον 21ο αιώνα. σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι χρειάζονται περισσότερος ΟΗΕ. Οπότε σας εύχομαι καλή τύχη. Θα είναι καλό όχι μόνο για τον ΟΗΕ αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο θέμα. Πρόκειται για την στρατηγική τη ευρωπαϊκή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω το λόγο, στο, το, την Προεδρία μάλλον, στον συνάδελφο. Τον συνάδελφο μου κύριο Πλένκοβιτς. Ο πρόεδρος Πλένκοβιτς. Ας συνεχίσουμε τι διαβουλεύσεις μας αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι στη σημερινή συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικών. Συνεχίζουμε με το υπαριθμό 9 της ημερησία διατάξεως που προβλέπει παρουσίαση της μελέτης προς μια νέα στρατηγική ασφαλείας ε, της Ευρώπης. Το μέρος αυτό της ενεργασίας μας γίνεται σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας την οποία εκπροσωπεί ο συνάδελφός μας κύριος Καν και καλωσορίζω τον κύριο Γιάνν Άντωνη που είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης. Θα έχετε δει ίσως στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία σας την μελέτη που είχε ανατεθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που συντάχθηκε σε συνεργασία με τις οργανώσεις Τσίτρι και Chatham House το Ινστιτούτο Στρατηγικών Ερευνών του Παρισιού. Είναι ε, πολύ επίκαιρη αυτή η συνάντηση και η συζήτησή μας, γιατί βρισκόμαστε λίγες ημέρες μόνο πριν από το ταξίδι της, μάλλον πριν από την παρουσίαση από την κυρία Μογκερίνη στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Αλλαγής των Αλλαγών στο Παγκόσμιο Περιβάλλον. Μια στρατηγική που έχει αρχίσει από το 2003, η οποία μετά αναθεωρήθηκε το 2008 και συνεχίζει τη συζήτηση στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πώς θα αντιμετωπιστεί το νέο πλαίσιο απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω. Το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο μπαίνει πραγματικά σε βάθος των προβλημάτων και έχει γίνει μετά από διαβουλεύσεις πανεπιστημιακών και άλλων αρμοδίων και γύρω από το θέμα της ε, στρατηγικής της ασφάλειας φαίνεται να δίνει συμβουλές και μεθοδολογικές και για την επιλογή, για τις πολιτικές επιλογές για το μέλλον της α, στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2005 και 2006 με θέματα όπως κυβερνοεπιθέσεις, υβριδική πόλεμη, τις σχέσεις με τη Ρωσία και με ορισμένου από του γειτονέ τη, θέματα τα οποία καλούμε θα λαμβάνουμε υπόψη όταν μελετούμε τη μελλοντική μα στρατηγική. Το άλλο θέμα είναι, σημειώνουμε εδώ, το τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως σημαντικός θεσμός. Περιλαμβάνουμε μια συζήτηση για την ε, στρατηγική και θέματα που έχουμε συζητήσει και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Βέβαια είναι μια στοχευμένη συζήτηση αυτή σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα θα προσφέρουμε και άλλες συνεισφορές και με την έκθεση της ΚΕΠΑ όπου περιλαμβάνεται και έκκληση για μια συντονισμένη προσέγγιση σε μια συνολική εξωτερική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καν να πει λίγα λόγια εκ μέρους της ΕΝΤΕ και μετά να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Είμαστε ιδιαίτερα, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για να ακούσουμε τις απόψεις σας για την νέα στρατηγική της Ένωσης. Όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το, του, το του 2013 ζήτησε από την ύπατη εκπρόσωπο να συντάξει έκθεση, την οποία θα υποβάλει άλλωστε η διάδοχό της σε λίγες ημέρες, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο πολύ θα άλλαζε ο κόσμος τους επόμενους μήνες. Δεν θα αναφερθώ και πάλι στην κρίση που αντιμετωπίζουμε, στις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε γύρω μας και γύρω από την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Είναι σημαντικό ωστόσο να τονιστεί ότι τα όσα συμβαίνουν και οι αντιδράσεις στα γεγονότα αυτά ή η έλλειψη αντιδράσεων κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τα όσα έχει επιτύχει μέχρι τώρα η παγκόσμια τάξη Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γίνουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις στο επίπεδο των θεσμικών οργάνων και αναμένουμε με ενδιαφέρον την περαιτέρω πορεία των προσπαθειών της εκ εκπροσώπου κ. Μογκερίνη. Οι πρόσφατες κρίσεις έχουν καταδείξει πόσο σημαντική είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή ενδέχεται να προκύψει. Και χρειάζεται μελέτη και των εξωτερικών και των εσωτερικών διαστάσεων. Στην υποεπιτροπή μας, ΣΕΝΤΕ, ασφαλώς και αποδίδουμε μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη σχετική συζήτηση. Η νέα στρατηγική της Ένωσης θα πρέπει κυρίως να προσφέρει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το πού θέλει να βρεθεί η Ευρώπη στον κόσμο και πώς θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια και εντός και εκτός των συνόρων της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο προστάσιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει από την διαχείριση των κρίσεων, την πολιτική ανάπτυξη διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλά χωρίς ένα συγκεκριμένο στρατηγικό όραμα, η χρήση των εργαλείων αυτών δεν μπορεί να αποδώσει τα βέλτιστα αποτέλεσματα. Σας ευχαριστώ που είστε παρόν κύριε Άντωνη και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας. Ο πρόεδρος Πλένκοβιτς, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Άντωνη, ο οποίος είναι άλλο εργάζεται τώρα στην Στοκχόλμη και θα μιλήσει βέβαια και για τα τρία θεσμικά όργανα που έχουν συμβάλει στην ε, εκπόνηση της εκθέσεως. Για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πρώτα για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στην σύνταξη της μελέτης που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για τα τρία και για τις τρεις οργανώσεις μας και για την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Δεν θα προσπαθήσω να συνοψίσω το περιεχόμενο του εγγράφου που φτάνει περίπου τις 100 σελίδες και δεν φτάνουν 15 λεπτά γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να έρθω σε μερικά από τα πιο ε, σημαντικά θέματα που περιλαμβάνει. Όταν αρχίσαμε, η απάντηση στην ερώτηση που έλεγε αν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση για μια νέα στρατηγική της ασφάλειας δεν ήταν αυτονόητη για μας η απάντηση στην ερώτηση αυτή. Αν εξετάσετε το έγγραφο του 2003 και το συμπλήρωμά του 2008, εξακολουθούν αυτά τα έγγραφα να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ωστόσο, μετά από τον προβληματισμό, καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ μιας νέας στρατηγικής προσέγγισης και ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να περιληφθεί τον μανδύα μιας νέας στρατηγικής της ασφάλειας. Έχει αλλάξει το παγκόσμιο περιβάλλον σε βάθος, τουλάχιστον σίγουρα από το 2003. Στην βάση των όσων βλέπουμε να γίνονται και μάλιστα πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δραματικές αλλαγές στα συστήματα ασφάλειας δεν μπορούν να αποκλείονται και πρέπει να προβλέπονται. Οι κρίσεις λοιπόν και οι προκλήσεις στην ασφάλεια που βλέπουμε θεωρούμε ότι δεν είναι του συνήθους είδους διότι βεβαίως ανά πάσα στιγμή εμφανίζονται κρίσεις, αλλά θίγουν κάποιες από τις πιο θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες έχει βασιστεί η στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί την αιτιολογία για μια νέα ματιά στο θέμα αυτό. Πέρα από αυτό, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει μέσα από ένα βαθύ μετασχηματισμό και με αλλαγές στα θεσμικά πλαίσια, διεύρυνση με την συμμετοχή νέων χωρών μελών που άλλαξαν σε βάθος την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μια συζήτηση για το αν θα πρέπει ενδεχομένως να σκεφτούμε μάλλον μια υποχώρηση μέσα στα όρια μας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες νομίζομαι ότι δικαιολογούν την έναρξη μιας νέας συζήτησης. Φύξαμε με λίγα λόγια τα όσα περιλαμβάνονται στο τμήμα 2 της έκθεσης που αναφέρεται στις απειλές. Όπως είπα, η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα αναπτύξω εν λεπτομερία. Ε, περιλαμβάνει τις διάφορες απειλές, είτε αυτές είναι άμεσες θανάσιμες απειλές, θανατηφόρες απόπειρες, απόπειρες σε βάρος της ζωής και της περιουσίας και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλές σε αυτό που λέμε τον τρόπο ζωής τον οποίο έχουμε συνηθίσει που μπορεί να είναι και εσωτερικές απειλές που απειλούν την ίδια την κοινωνική συνοχή ζημιές στην ίδια την οικονομία, στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διείσδυση μέσα στις κοινωνίες από την οργανωμένη εγκληματικότητα, όλες αυτές οι απειλές λοιπόν μια τρίτη ομάδα απειλών είναι απειλές κατά ευρωπαϊκών συμφερόντων σε άλλα μέρη του κόσμου. Καμιά φορά άμεσες, για παράδειγμα απαγωγές Ευρωπαίων πολιτών σε περιοχές κρίσεων, απειλές κατά εξωτερικών επενδύσεων που έχουν κάνει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, υπονομεύουν όμως και την ίδια την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσω συγκρούσεων που καταστρέφουν υποδομές, που καταστρέφουν την πρόοδο στους χώρους της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, αλλά και άλλοι παράγοντες. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα που είναι ο ιός έμπολα στην Δυτική Αφρική, που μέσα σε λίγους μήνες κατέστρεψε, ανέτρεψε πρόοδο δεκαετιών. Τέλος, απειλές σε ευρωπαϊκούς, κατά ευρωπαϊκών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται σε ένα σύστημα κανόνων και πολυμερούς αντιμετώπισης και εδώ μπορεί να υπάρξει απειλή σε βασικές ευρωπαϊκές αρχές οι οποίες εφόσον εφαρμόζονται είναι ασφαλώς προς όφελός μας σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν τέσσερις διαφορετικές, τέσσερα διαφορετικά ίδια απειλών, αλλά η ισορροπία μεταξύ τους αλλάζει επίσης. Ένα από τα συμπεράσματα της ε, εκθέσεως είναι ότι η πρώτη ομάδα απειλών, οι άμεσες απειλές δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνουν περισσότερη βαρύτητα τώρα από ότι μέσα στην προηγούμενη δεκαετία. Αυτό βασίζεται και στην ανάλυση που κάνουμε των τάσεων των απειλών μετά από μια δεκαετία θετικών εξελίξεων με την έννοια ότι μειώνεται ο αριθμός των συγκρούσεων τα δεδομένα που συλλέγουμε και αναλύουμε τώρα δείχνουν ότι τα τελευταία τρία χρόνια περνούμε ένα σημείο καμπής και προχωρούμε τώρα σε μια αρνητική εξέλιξη. Βλέπουμε αύξηση των συγκρούσεων και βλέπουμε και αύξηση των εντάσεων των συγκρούσεων. Είναι νωρί ακόμα για να μιλήσει κανείς για μια συνολικότερη τάση. Όμω τρία χρόνια τώρα τα δεδομένα που συλλέγουμε δείχνουν ότι δεν πάμε προς τη κατεύθυνση. Δεύτερο, οι απαιτήσει διασφάλισης και των χωρών τη Ενώσης και των στενών μας εταίρων. Εφόσον ληφθούν εκ παραλίλου με τις αυξημένες απαιτήσει ειρηνευτικών παρεμβάσεων και εκτός Ευρώπης, ιδίως στην Αφρική δε, πάλι τα δεδομένα που συλλέγουμε και δημοσιεύουμε δείχνουν ότι τώρα για τρίτη συνεχή χρονιά ο αριθμός των παρεμβάσεων αυτών έχει αυξηθεί. Υπάρχει λοιπόν αυξημένη αυξημένες απαιτήσει απέναντι στους πόρους που διαθέτουμε και εντός Ευρώπης και εκτός. Εκτιμώντας την ισορροπία αυτών των απειλών δείχνουν, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Πολλές από τις απειλές που έχουμε εντοπίσει και δεν μας εκπλήσει αυτό οφείλουν να θεωρηθούν ως συστημικές. Δεν παραμένουν μέσα στις παραμέτρους των εθνικών συνόρων, χρειάζονται συνδυασμό του ιδιωτικού και του δημόσιου παράγοντα. Πρόκειται για συστημικές απειλές λοιπόν, οι οποίες ξεπερνούν τις ικανότητες μιας μεμονωμένης χώρας μέλους, ακόμα και αν είναι από τις μεγαλύτερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί είναι σημαντικοί λόγοι για να αντιμετωπιστεί, που συνηγορούν υπέρ της αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού στο ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο καθίσταται αναγκαίο. Εάν επιστρέψουμε στο τελικό, στο τμήμα 3 της εκθέσεώς μας, Πάλι το τμήμα αυτό είναι αρκετά μακροσκελές. Εδώ επιθυμώ να σας επισημάνω ένα πράγμα. Θα πω για τα πιο όριμα φρούτα, τους πιο όριμους καρπούς, αν μπορώ να το πω έτσι. Πράγματα που μπορεί να γίνουν με σχετικά χαμηλό κόστος, χωρίς ανάγκη σημαντικών σε βάθος αλλαγών στο παρόν περιβάλλον και βασίζονται στην δουλειά που έχει ήδη γίνει για να αυξηθεί η συνοχή με πρακτικό τρόπο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών, κυρίως συγκέντρωση των στοιχείων του ενεργητικού που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε περιοχές συγκρούσεων, προώθηση του συλλογικού σχεδιασμού, εφαρμογή με κοινέ πρωτοβουλίες και διασφάλιση του ότι θα γίνεται ανάλυση των συγκρούσεων και ανάλυση των απειλών σε όλες τις χώρες και όχι μοναχά σε χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Κάτι το οποίο ε, έχει τονιστεί ως ανάγκη στην Ουκρανία, όπου βλέπουμε την ανάγκη να γίνεται ανάλυση συγκρούσεων και σε χώρες που δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αν προχωρήσουμε τώρα στο τελικό τμήμα της εκθέσεως, όπου μιλούμε για τις συστάσεις, για το τι πρέπει να γίνει δηλαδή με κάπως πιο φιλόδοξο τρόπο, Εκεί εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μας απασχολήσει η διαδικασία, δηλαδή το πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια στρατηγική ασφαλείας, καθώς και ποιοι πρέπει να είναι οι αντικειμενικοί στόχοι της. Οι βασικοί στόχοι και η μεθοδολογία εργασίας εξηγούνται στο τελευταίο τμήμα της εκθέσεως. Εξηγείται εκεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλει να εξηγήσει το ρόλο της στο κοινό στην κοινή γνώμη να προσφέρει και κατευθυντήρες γραμμές καθοδήγηση για το πώς θα πρέπει να δρουν τα μέλη για παράδειγμα των διαφόρων θεσμών, πώς θα συμβάλλουν για να επιτευχθεί ένας ευρύτερος στόχος, να δοθεί και ενίσχυση στους εταίρους μας απαντοχού του κόσμου να κατανοήσουν πώς μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αμοιβαίο όφελος, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και εκτός Ένωσης λαμβάνονται υπόψη οι οπτικές γωνιές των χωρών μελών, των κοινοβουλίων και της κοινή γνώμη και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργηθεί και η συνένεση που απαιτείται. Αυτό βέβαια σε αντίθεση με τον τρόπο που είχε συνταχθεί το έγγραφο του 2003. Μια διαδικασία συμπερίληψης θεωρούμε ότι θα παραγάγει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο ωστόσο να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα πολύ συμπιεσμένο χρονικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια διαδικασία που φαίνεται να κινείται μέσα σε κύκλους περίπου δεκαετίας. Να συνταχθεί ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί να ισχύει και σε μια δεκαετία από σήμερα είναι και χρήσιμο και αναγκαίο να δαπανηθεί ο σχετικός χρόνος καλύτερα παρά να μπουν κάποιες τεχνητές προθεσμίες του εξαμήνου για παράδειγμα. Εφόσον πρόκειται να το κάνετε μια φορά ανά δεκαετία, καλύτερα να είναι σωστά. Η βασική προσέγγιση, όπως εξήγησα, είναι ευρύτατο το φάσμα των διαφόρων τύπων απειλών που οφείλουν να ληφθούν υπόψη στην έρευνα και βεβαίως και μια μακροπρόθεσμη προοπτική, καθώς και στόχευση και στις άμεσες απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα αντιμετωπίσει βεβαίως σοκ, αναταράξεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αυτή λοιπόν στιγμή γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν οι αναταράξεις αυτές και δεν μπορούμε να πούμε ακρίβεια τι θα είναι αυτές και πού θα είναι αυτές. Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα πρέπει να είναι η δημιουργία ανθεκτικότητας ως βασικό, ως στοιχείο κλειδί της στρατηγικής αυτής. Να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και να αντιμετωπίσουμε τα υπερχόμενα γεγονότα να τα προβλέπουμε και να προβλέπουμε και τις επιπτώσεις που θα έχουν στον τρόπο ζωής μας και στη ζωή των πολιτών. Τρίτο στοιχείο που θα πρέπει να είναι βασικό, να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποσυρθεί από τα παγκόσμια πράγματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ισχύσει μια ρεαλιστική άποψη σχετικά με το πού μπορεί να συμβάλλει επικοδομητικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιου είδους παρεμβάσεις θα αποφέρουν το μέγιστο όφελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει σημαντικό παράγοντα σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όμω να λύσει όλα τα προβλήματα σε όλε τι περιοχέ του κόσμου. Τέλο ω ένα από τα στοιχεία τη βασική προσέγγιση, απομόνωση δηλαδή και οριοθέτηση των τομέων εκείνων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει ως μοναδικός παράγοντας. Κανένας δηλαδή άλλος δεν μπορεί να προσφέρει τόσα ή τόσο καλά. Ένας τομέας όπου είναι ουσιώδης και πρέπει να στοχεύσουμε σε αυτόν είναι η κατανόηση και αντιμετώπιση της διασύνδεσης μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Στον τομέα αυτό έχει ήδη παίξει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατανόηση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Μπορώ ε, ε, ε, Έχει μεγάλη τεχνογνωσία βεβαίως και μπορεί και να κάνει και τις ίδιες διαδικασίες τις πιο αποτελεσματικές και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία. Μια αξιολόγηση των διαφόρων εταιρικών σχέσεων. Θα είμαι ειλικρινής, θα πω σε αυτό το τομέα δεν πετύχαμε πλήρη συμφωνία όσοι ετοιμάσαμε την έκθεση. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί μέσω εταιρικών σχέσεων αλλά πρέπει να έχουμε σαφή εικόνα του τι εννοούμε μέσω στρατηγικού εταίρου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, είπα, είναι προφανής περίπτωση όπου η σχέση μας είναι τόσο στενή που δεν έχει σημασία να αποκαλειται στρατηγική εταιρική σχέση, θα έχει τα χαρακτηριστικά της όμως. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου βλέπει κανείς, όπου υπάρχει η προοπτική η στρατηγική συνεργασία, στενή συνεργασία με ένα σταθερό εταίρο με άλλα λόγια, αλλά δεν είναι σαφές ποια θα είναι η ουσία των υφισταμένων ε, στρατηγικων εταιρικών σχέσεων. Με χώρες πραγματικά χρειάζεται να εστιάζεσαι επί διαφόρων σημείων όπως της Νοτιού Ασίας, Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα κλπ. Σε ποιο βαθμό δηλαδή αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση που δηλώνουμε έχει κάποιο νόημα. Και υπάρχουν χώρε με τι οποίε είπαμε ότι έχουμε στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει και πιθανότατα δεν έπρεπε να έχουμε κατά παρελθόν και σίγουρα δεν έχουμε τώρα, όπω είναι η Ρωσία το προφανέστατο παράδειγμα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι εννοούμε με την έννοια στρατηγικό εταίρο, να εστιαστούμε επί τη ουσία και περιεχομένου τη στρατηγική εταιρική σχέση. Αυτό είναι ένα πολύ απαραίτητο στοιχείο. Επόμενο σημείο, περιφερειακέ προκλήσει αφορά την ασφάλεια. Διαφαίνεται σαφώ από την έκθεση ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υπάρχει μια παγκόσμια τάξη δυνάμει κανόνων, υπάρχουν πολλέ ε, προκλήσει στη γειτονιά μα που απαιτούν την προσοχή μα. Και αυτό δεν μπορεί να βληθεί και δεν μπορεί να προσεγγιστεί σταδιακά. Πρέπει να εστιαστούμε επί προκλήσεων για την περιφερειακή ασφάλεια και αυτό είναι επιτακτική ανάγκη. Και τέλος να εστιαστούμε επί των εγκαρσίων προκλήσεων. Όπως προανέφερα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη βασική της προσέγγιση, να είναι ανοιχτή, να συμμετέχει στα παγκόσμια τεκτενόμενα, είναι προς όφελός μας, αλλά δημιουργεί και κάποια σημεία δυναμίας. Γινόμαστε ευάλωτοι. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε θετικέ ροέ, είτε είναι άνθρωποι, ιδέε, χρηματοδότηση, χρηματοπιστικά, στατικικά αγαθά, αλλά αυτά μπορούν να αποτελούν και τα σημεία. Δημιουργούν ε, διόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, διάφοροι ε, άνθρωποι που έχουν κακές διαθέσεις. Είναι περίπλοκο το θέμα, πολύ περίπλοκο, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό σε οποιοδήποτε επίπεδο. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση εγκαρσίων προσεγγίσεων. Από τη φύση του αυτός ο τομέας μπορεί να βοηθήσει να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ε, προστασία για τη δική της ασφάλεια αλλά όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτά ήθελα να αναφέρω, να θίξω από την προσέγγιση. Περίπου 100 σελίδες περιέχει, θα ήταν πολύ κουραστικό να συνοψίσω κάθε σημείο ή να διαβάσω την έκθεση. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντωνη. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας, ούτως ώστε όλοι οι συνάδελφοι που θέλουν να συμμετάσχουν να μπορούν να το κάνουν. Αν μου το ζητήσουν, έχω 6 συναδέλφους για την ώρα που είναι στον κατάλογο, 7 θα προσπαθήσω να δώσω 3 λεπτά στον καθένα το πολύ, νομίζω ότι αρκεί. Ούτως ώστε να απαντήσει και ο κύριος Άντωνη. Η κυρία Καλνιέτε έχει το λόγο εκ μέρους ε, του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ε, διεξοδικότατη έκθεση και η παρουσίαση. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια καλή βάση για την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων και για την Επίτροπο την κυρία Μογκερίνη στην προσπάθεια που καταβάλουν να δημιουργήσουν μια νέα στρατηγική ασφαλείας για την ε, Ευρώπη Υπάρχουν αρκετά σχόλια στα οποία θα επιθυμούσα να προβώ. Το πρώτο σχόλιο σχετίζεται με τους γείτονές μας. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να αποφύγουμε το κεντρικό ζήτημα το οποίο χρήζει απαντήσεως Τι είδου σχέσει θέλουμε, τι είδου μέλλον θέλουμε με τους γειτονέ μας. Θα μιλήσω λετωνικά, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, τρεις από τις γειτονικέ μας χώρες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι αυτό δείχνει κάποια ποιότητα των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσφέρουμε στους γείτονές μας και άλλους τρόπους συνεργασίας, ούτως ώστε οι γείτονές μας αυτοί να κινηθούν σε πλαίσια διαλειτουργικότητας. Να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ γειτόνων και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να το πούμε. Αναφέρομαι εδώ στην ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας στο Στασβούργο όσον αφορά τη στρατηγική ασφαλείας για τον εύξηνο πόντο, όπου στο άρθρο 16 δεν θέλαμε να γίνεται αναφορά στη συνεργασία μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ και της Γεωργίας και της Μολδαβίας και της Ουκρανίας Απ' την άλλη, νομίζω ότι η συνεργασία για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα όσον αφορά τη Γεωργία, η Γεωργία έλαβε υποσχέσεις που αφορούσαν το ενδεχόμενο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό έγινε Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες όσον αφορά τις απειλές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι θέσεις προτεραιοτήτων δεν θα είναι κάτι εύκολο, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μιλήσουμε για την κυβέρνοασφάλεια, τις σχετικές απειλές, μετά υποδομές, πυρηνικού σταθμούς παραγωγής ενέργειας, και τελευταίο τομέα η τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε όμως σημαντικότατη πτυχή που είναι η προπαγάνδα. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ευρωπαϊκούς λαούς από την μαζική πληροφόρηση και διάφορες εκστρατείες πλήσης εγκεφάλου. Ευχαριστώ πολύ Σάντρα. Ο συνάδελφος Μπαλτσίτης έχει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Θέλω όμως να αναφερθώ σε δύο πτυχές. Πρώτον, δεν αναφερθήκατε σε εσωτερικές προκλήσεις που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι μιλάμε για την αλληλεγγύη που σίγουρα αποτελεί τη βάση για όλες τις χώρες μέλη όμως από τα σημερινά γεγονότα βλέπουμε ότι όταν ψηφίζουμε τη μία την άλλη έκθεση είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν αναφερθήκατε σε έναν από τους κύριους παράγοντες που είναι το ενεργειακό. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε κατά της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενέργεια που εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα από τα έγγραφα κλειδί που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες. Και το έγγραφο αναφέρει διάφορες πτυχές για τις οποίες οι χώρες μέλη δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα εξαιτίας των οικονομικών τους συμφερόντων. Σχέσεις με τη Ρωσία για παράδειγμα. Εσείς αναφερθήκατε στη συνοχή στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάντα ένας παγκόσμιος παίχτης, όμως από την τρέχουσα κατάσταση είναι σαφές ότι είμαστε διχασμένοι και αν δεν μπορέσουμε να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις επιμέρους χώρες μέλη, μπορεί να αποδυναμωθούμε ακόμα περισσότερο ως παγκόσμιος παίκτης. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια πρέπει να αναλύει και αυτά τα στοιχεία. Τέλος, όσον αφορά τη συνοχή στη δράση μας. Κάθε χώρα μέλος έχει εκλογές κάποια στιγμή και προκειμένου να εφαρμοστούν κάποια στοιχεία της στρατηγικής ε, πρέπει να προχωρήσουμε σε δράσεις που δεν είναι πάντα τόσο δημοφιλείς. Υπάρχει το δημογραφικό ζήτημα βέβαια, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη στρατηγική μας και στις εξωτερικές μας δράσεις. Ευχαριστούμε κύριε Μπουλσίτης. Ο κύριος Βανόρντεν τώρα, από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Άντωνη για την παρουσίασή σας. Δεν είχα την ευκαιρία να τη διαβάσω διεξοδικά λίγο. Η εντολή σας ήταν προφανώς να βρείτε κάποιο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους αυτούς τους τομείς. Βασικά έναν πιο προθυμένο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως προϋποθέτει κοινά συμφέροντα που ίσως να υπάρχουν βέβαια σε κάποιους χώρους, αλλά σίγουρα όχι σε όλους. Δεν αφισβητείτε καθόλου τις υποθέσεις αυτές, τις προϋποθέσεις αυτές, οπότε να ρωτιέμαι σε τι βαθμό έχετε συζητήσει την αναζωγόνηση του ΝΑΤΟ, αναφέρεστε στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι σε αυτά τα πλαίσια. Η απάντηση στις διάφορες απειλείς που αναφέρεται επόκειται στις εθνικές μας κυβερνήσεις. Ε, φυσικά κάπου χρειαζόμαστε συμμάχους όπου υπάρχει το διασυνοριακό που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όμως τα περισσότερα προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις κυβερνήσεις μας. Οπότε η ερώτησή μου είναι, τι χρησιμότητα ε, μπορεί να υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέγαμε κάποια μη στρατιωτικά μέσα αναφερθήκατε την αναπτυξιακή, στην αναπτυξιακή βοήθεια, ναι, αλλά και πάλι σε τι βαθμό η χρήση των μέσων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετούν τους σωστούς στόχους. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν ε, και ένα που έχω στο μυαλό μου τώρα είναι η μόχλευση που θα έπρεπε να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση της Παλαιστινικής Αρχής, προκειμένου να λυθεί το ειρηνευτικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή. Στο κάτω-κάτω είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να έχουμε αυτήν την πολιτική μόχλευση προκειμένου να βρεθεί πιο εύκολα λύση. Σε τι βαθμό λοιπόν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τις δυσκολίες. Το θέμα της μετανάστευσης, μεταναστευτική πολιτική. Να, άλλο παράδειγμα. Σε τι βαθμό η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί οι άλλες βοηθούν. Αντίθετα, κάποιες κάνουν πιο έντονο το πρόβλημα αντί να το ξεπερνούν. Και όταν μιλάτε για τους στόχους, ο πρώτος που αναφέρατε ήταν η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόθεση της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος στόχος θα έπρεπε να είναι πώς θα ξεπεράσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Πού πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της και την προσοχή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα επίσης να ακούσω από εσά ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να δαπανούν περισσότερα στην άμυνα. Ευχαριστώ. Συναδελφοί, όχι πάνω από τρία λεπτά για να προλάβουμε να έχουμε και συζήτηση και απαντήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τους συντάκτες της έκθεσης αυτής. Η ευρωπαϊκή μας ε, αυτή η στρατηγική ασφάλειας χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Είμαστε μπροστά σε μια νέα στρατηγική λοιπόν και το ζήτημα είναι το κατά πόσο επιθυμούμε να έχουμε μια καλή νέα στρατηγική. Η πρώτη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να ορίσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Να δούμε τις σχέσεις μας με όλες τις αμερικανικές χώρες. Υπάρχουν δύο ζητήματα που δεν είναι σαφή και έχουν να κάνουν ακριβώς με τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή σχέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Έπειτα μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Στο ΝΑΤΟ ένας πυλώνας υπάρχει. Και αυτός είναι Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε. Και υπάρχουν και 21 μικροί πυλώνες από δίπλα. Είναι ψευδέστηση λοιπόν να μιλάμε για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα μέσα στο ΝΑΤΟ. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να δρά συμπληρωματικά με τον ΝΑΤΟ. Κάτι παράδοξο, αφού γνωρίζουμε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ επίσης. Άρα συμπληρωματική πολιτική στον εαυτό τους αυτό είναι το παράδοξο. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή. Υπάρχει δυνατότητα σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΝΑΤΟ θα μπορούσε να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα μέσα στα πλαίσια της νέας στρατηγικής. Η κυρία Λούζιν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εσείς κύριε Άντωνη, μιλήσατε για σενάρια απειλών και μεταξύ αυτών αναφέρατε και το οργανωμένο έγκλημα. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι καθαρά πτυχή εσωτερικής πολιτικής. Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι υπόθεση της αστυνομίας. Βλέπω εδώ να ακολουθείτε μια, α, μια πορεία περιορισμού της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας και ενδεχομένως μια σύγχυση στρατιωτικών και αστυνομικών καθηκόντων. Κάτι το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί και με κάποιες συγκεκριμένες ερμηνείες της ρήτρα αλληλεγγύης. Γι' αυτό και η ερώτησή μου. Θεωρείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος σύγχυσης στρατιωτικών και αστυνομικών καθηκόντων και κατά πόσο θεωρείται αυτό ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα δημοκρατικής διάκρισης των λειτουργιών. Και έχω και μια ερώτηση για τον χώρο γειτονίας. Στη μελέτη ζητείται κατ' η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στον χώρο της γειτονίας της. Εκεί είπαν και διάφορα οι συναδελφοί μου, ως λογική συνέπεια του ρόλου της Ρωσίας, που εμφανίζεται βέβαια πάντοτε μονομερός σαν μια ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης. Η ερώτηση λοιπόν προς εσάς στο σχετικό κεφάλαιο είναι αρκετά ασαφής η περιγραφή. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι επιπτώσεις από την στρατιωτική πλευρά. Και η συγκεκριμένη με ερώτηση είναι εάν στην συμπερίληψη των συμφωνιών ε, ε, πολιτικής γειτονίας, η συμπερίληψη των στρατιωτικών πτυχών μπορεί να θεωρηθεί ως λύση κάποιου προβλήματος. Πώς το ερμηνεύεται αυτό. Και έχω και μια ερώτηση τώρα, τέλος, για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Αναφέρομαι πάντα σε αριθμούς του Ινστιτούτου Σύπρη, όπου εμφανίζεται η σημαντική μείωση των εξοπλιστικών δαπανών ως απειλή. Αν όμως ερμηνεύω σωστά τους αριθμούς του Σύπρη, δεν μπορεί να μιλεί κανείς για σημαντική μείωση των εξοπλιστικών δαπανών. Αν πάρω για παράδειγμα τους αριθμούς του 2.270 εκατομμύρια ευρώ, ε, δισεκατομμύρια ευρώ, μέχρι το 2013 που είναι λίγο παραπάνω 279 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν βρίσκω να υπάρχει καμιά σημαντική μείωση. Πώς εξηγείτε, πώς ερμηνεύετε τα νούμερα αυτά εσείς οι ίδιος. Ευχαριστώ. Ο κ. Κάρβερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλουμε πιο φιλόδοξη πολιτική ασφάλεια. Περισσότερη πτυχή Ευρωπαϊκής Ενώσεως. εξελέγει στο Κοινοβούλιο πέρσι. Και όλο και περισσότερο Ευρώπη και λιγότερο κράτη-μέλη βλέπουμε. Είναι ηρωνικό αυτό, διότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα στη χώρα μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και γίνεται αναθεώρηση πολιτικών ασφαλείας σε πολλά κράτη-μέλη. Και είναι ηρωνικό που η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ενώσης μπορεί να είναι ει βάρο της περιφερειακής και ενδεχομένω παγκοσμία ασφαλείας. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στου πυλώνε του ΝΑΤΟ. Τον είπα, τον ευρωπαϊκό πυλώνα, ποια είναι η απόψή σα. Κατά την άποψή μου, το ΝΑΤΟ δεν έχει πυλώνε Αποτελείται από κυρίαρχα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Και τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να αποφασίζουν σε ποιους τομείς, σε ποιες περιοχές θέλουν να επέμβουν για τα εθνικά του συμφέροντα. Εγώ δεν ανήκω ότι ανήκω εδώ και λέω όπως θέλετε να αναπτύξετε μια στρατηγική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θεωρούμε ότι αυτό είναι εις βάρος των κρατών μελών. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Ευχαριστώ. Τόνι Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σημαντική έρευνα. Πέρασαν 12 χρόνια από την περασμένη στρατηγική ασφαλείας. Και όπως είπατε ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο ευημερής, πιο ασφαλής και πιο ελεύθερη όπως ήταν πριν από 12 χρόνια. Τώρα η διεθνής τάξης έχει παραβιαστεί. Έχουν καταρρεύσει κάποια σημεία που αφορούν την ασφάλεια, χρειάζεται σαφές στατηγικό όραμα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά τη νέα κατάσταση και τις αντιδράσεις που απαιτούνται. Λείπει και η ενότητα. Ανησυχώ κάπως. Ανησυχώ λόγω των προτάσεών σας στη σελίδα 44. Πώς να αντιδράσουμε στη Νέα Ρωσία. Λέει ότι έχει πιο επιθετική εξωτερική πολιτική η Ρωσία και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό είναι άλλος ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και καταλήγει ότι η νέα πολιτική ασφαλείας πρέπει να κατανοεί το στρατηγικό όραμα της Ρωσίας και να υπάρχει και ένα αντίθετο από την πλευρά μας προοδευτικό στατικικό όραμα. Θεωρητική αυτή η πρόταση. Δεν ξέρω αν έχει πρακτική αξία. Αμφιβάλλω. Προσπαθούμε να βρούμε απάντηση σε αυτό στο ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας που αφορούσε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ρωσίας. Εκτιμώ τα μάλα τις εταιρικές σχέσεις. Μας χρειάζονται αλλά χρειάζεται καλύτερος και ακριβέστερος ορισμός της ενίας εταιρική σχέση. Κυρίως όσον αφορά την τεχνολογία το κυβερνοχώρο, τις απειλές για τις ζωτικές υποδομές. Έτσι η παρουσίαση θα είναι πολύ πιστική και αναλυτική. Πρέπει να τονίσουμε τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ παραπάνω αυτό αναφέρει. Έχω αμφιβολίες όσον αφορά το τμήμα για το Ιράν. Δεν συμφωνώ με τα συμπεράσματα. Δηλαδή, ότι οι διαπραγματεύσεις άλλαξαν την κατάσταση και ότι πάγωσε η πυρηνική έρευνα και τα διάφορα προγράμματα τα σχετικά για τα πυρηνικά στο Ιράν. Δεν έχουμε δει τις ενδείξεις. Ανοιχτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πραγματικά τα όσα συμβαίνουν εντός της χώρας, εντός του Ιράν. Ευχαριστώ Τούνε. Μπορείς Σόλιτα. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια έχω. Ο κύριος Ζάλα, συγγνώμη, για τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Καλό το ότι ο κύριος Άντωνη αναφέρθηκε σε αυτό. είχαμε μια όχι πολύ θετική εμπειρία όσον αφορά τον επεκτατισμό του κυρίου Πούτιν. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε λοιπόν το όλο πρόβλημα. Σημαντικότατο κατά την άποψή μου. Στην έννοια αυτή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ιδέες μας και τις αξίες μας. Δεν είναι μια θεωρητική κατηγορία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πραγματικά εργαλεία για τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις όχι μόνο με τις χώρες που ενστερνίζονται τις ίδιες αξίες, αλλά να διαδώσουμε τις ιδέες μας και τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όταν αναφέρθηκα στη Νότια Αφρική, για την υποσαχάρια Αφρική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και άλλες χώρες στην νότια, στα νότια της Αφρικανικής Υπήρου. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις χώρες από τη Βόρεια Αφρική, από την Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, λέει ο μιλήτης, πρέπει να ανανεωθεί, για να γίνει αυτό, να ανανεωθεί η έννοια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Μετά, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θεωρούμε ότι είναι κάτι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι που μας χρειάζεται. Χρειαζόμαστε δική μας ευρωπαϊκή στρατηγική για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ ε, σαν φορέας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας πυλώνας μια, ενός οργανισμός με έναν πυλώνα. Οι γειτονικέ χώρες της Ρωσίας, οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, οι άλλες ανατολικές χώρες, όταν ζητούν βοήθεια, ζητούν στρατούς και όπλα των ήπα Δεν ζητούν τα όπλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, ούτε καν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι στρατηγική πρόκληση για μας. Πρέπει να επανεξετάσουμε τη νέα ε, κατάσταση που δημιουργείται λόγω της τάσης της ε, Ρωσίας. Ευχαριστώ κύριε Ζάλα. Συνάδελφε Γιούρεκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την μελέτη, πολύ χρήσιμη, που έχετε υποβάλει κύριε Άντωνη. Έχετε θέσει πολλά σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικό επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με υπεύθυνο τρόπο στη θέσπιση της μελλοντικής στρατηγικής. Ωστόσο σημαντική είναι και η αλληλεγγύη απέναντι στις χώρες εκείνες των οποίων απειλείται η εδαφική ακαιρεότητα. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φανεί υπεύθυνη, να, να χειριστεί υπεύθυνα τα θέματα αυτά και των χωρών που βρίσκονται στην άμεση γειτονία μας. Αναλαμβάνει παρεμβάσεις σε μακρινά μέρη του κόσμου, αλλά θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στα πιο σημαντικά μας καθήκοντα που είναι αυτά. Κάθε μήνα που συνεχίζεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και η δική μας ασφάλεια απειλείται περισσότερο. Οι εντάσεις συνεχίζονται, όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, τόσο περισσότερο καθίσταται σαφές ότι η βία μέσα στον 21ο αιώνα ξαναγίνεται εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η πραγματική απειλή κατά της παγκόσμιας τάξεως. εάν κινηθεί απειλητικά η Ρωσία απέναντι μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Και η επιλογή θα είναι είτε πόλεμος, είτε θα καταστρέψουμε τότε την βάση της συλλογική μας ασφάλειας που αποτελεί το ΝΑΤΟ. Αντιμετωπίζουμε πλήθος συγκρούσεων εδαφικών, ε, θρησκευτικών, πολιτιστικών και ούτω καθεξής. Σε όλες αυτές τις ε, συγκρούσεις ένα ρόλο παίζουν κυβερνήσεις που καμιά φορά αποτελούν απειλή για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων και την θέτουν σε κίνδυνο. Τέλος, κάτι το οποίο θεωρώ ότι οφείλω να επισημάνω. Εάν στρέψουμε τα βλέμματα προς το μέλλον και διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος κλιμακώσεως στην Ουκρανία, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να αποκαταστήσουμε την περιφερειακή σταθερότητα στην περιοχή αυτή του κόσμου. Αυτό θα είναι το μέτρο για την εξωτερική μας πολιτική. Το πώς θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε σε τέτοιες εξελίξεις. Επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμη ότι η καλύτερη απάντηση εκ μέρους μας θα είναι να ανοίξουμε τις οδούς συνεργασίας με την Γεωργία και να ενισχύσουμε τη δυνατότητα, την αμυντική ικανότητα των βαλτικών χωρών. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για οργανισμό που είναι το θεμέλιο της δυνατότητας αντίστασης των χωρών μας. Είναι ο πρώτος θεμέλιος δίθος και αυτόν πρέπει να στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Κόζε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο έχει αποτύχει η πολιτική ασφάλειας μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση; Μα βέβαια, αφού έχουμε πόλεμο, εννοείται, έχουμε πόλεμο. Το λέγαμε το 2008. Μετά αναγνωρίσαμε το κοσυφοπέδιο, διεύρυνση του ΝΑΤΟ, οι δυνάμεις ε, βρεκανές θέσεις. Δεν είναι ψυχρός πόλεμος, πολύ θερμός θα έλεγα. Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος με αυτά που ανακοινώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τη δυνατότητα να αναπτύξουν ε, μαχητές και όπλα στις ε, βαλτικές χώρες και στην Πολωνία και την ε, Ρουμανία. Και η Ρωσία είπε ότι τότε θα απαντήσει με τα δικά της, ε, τα MRM στη, στο Καλίνικρατ, που μπορούν να έχουν πυρηνικές κεφαλές. Πώς θα πετύχουμε την ειρήνη έτσι. Η Ρωσία λέει ότι και στη Λευκορωσία θα στείλει αεροπλάνα. Μιλάμε για προπαγάνδα. Ε, είμαι δημοσιογράφος και ξέρω ότι είναι προπαγάνδα. Και εμείς κάνουμε προπαγάνδα και άλλοι κάνουν προπαγάνδα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το ότι το CNN που το βλέπουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι ενώ 300 εκατομμύρια βλέπουν τα ρωσικά μέση ενημέρωση. Το είπε η Χίλερη Κλίντον. Υβριδική πόλεμη. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, πόλεμη τέταρτης γενιάς από τις ΗΠΑ. Ποιος το έκανε πρώτο. Ε, είναι το θέμα ε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό η κότα. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι περισσότερο Ευρώπη και λιγότερο Ε για να μην καταλήξουμε στην αποτυχία της στρατηγικής μας ασφάλειας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καν πρώτος να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε Καν. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Για μένα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Το πρώτο είναι οι συζητήσει για την τρομοκρατία και άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την τρομοκρατία και την αντιτρομοκρατία. Αυτό που λέτε είναι ότι υπάρχει μείωση στις επιθέσεις και στις συλλήψεις. Θα συνεχιστεί η τάση αυτή. Και τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να μειωθεί ο ρυθμός ακόμα πιο έντονα. Δεύτερη ερώτηση. για τα drones, τα μη επαδρομένα αεροσκάφη και τη μη στρατιωτική χρήση τους. Οι Πολωνοί πώς βλέπουν το θέμα της ασφάλειας από τα αεροσκάφη αυτά. Πόσο πρέπει να λειτουργούν ακόμη και τα στρατιωτικά πρέπει να ακολουθούν κάποιο διεθνή κανόνα. Και έπειτα η απειλή από αυτήν την ε, τεχνολογία πέφτει και σε μη κρατικού ε, παίκτες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ερώτηση από μένα γιατί και εγώ προσπάθησα έτσι κάπως γρήγορα να διαβάσω την έκθεση αυτή. Δεν είπατε πολλά για τον προπολογισμό, για τα κονδύλια, εξωτερική πολιτική. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για το 2016 που θέλουμε να υπάρξει αύξηση πληρωμών. Αυτό προβλέπει η πρόταση. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Γιατί νομίζω ότι και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία της εξωτερικής μας πολιτικής. Ευχαριστώ. Τώρα, έχετε 10-12 λεπτά για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ. Δεν θα απαντήσω κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο βασικό πνεύμα των ερωτήσεων, στο βαθμό που δίναμε. Ας ξεκινήσουμε με το κατά πόσο ζητά περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη η έκθεση. Τι λέει η έκθεση ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των ήδη τεκτενωμένων. Όχι να επεκτείνουμε, να βελτιστοποιήσουμε αυτά που ήδη κάνουμε. Να εντοπίσουμε τους τομείς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία και να το αποδείξει. Αυτό λέει η έκθεση και τίποτα άλλο. Αν στραφούμε τώρα στις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ και τα συναφή αν απομακρυνθούμε λίγο από το θέμα, τι έγινε το τελευταίο χρόνο, τελευταία δύο χρόνια, είδαμε τα μάτια μας το πώς η συλλογική ασφάλεια προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, τώρα αρχίζει και μειώνεται η ασφάλεια. Έχουμε δημιουργήσει θεσμούς, διαδικασίες και από πολιτική κρίση σε τέσσερις μήνες περάσαμε σε σύγκρουση, σε μια σημαντική ευρωπαϊκή χώρα κάποιο παρουσιάστηκαν σαν επιτυχίες της τάξης όσον αφορά την ασφάλεια, αποστατικοποίηση της ευρωπαϊκής ασφαλείας από τα φρικτά επίπεδα που φτάσαμε στο ψυχρό πόλεμο, τώρα όλα αυτά παρουσιάζονται φάλματα και αδυναμίες. Βασικό ερώτημα. Πώς μπορούμε να επανέλθουμε πίσω στο μονοπάτι να δημιουργήσουμε συλλογική ευρωπαϊκή ασφάλεια Μακροπρόθεσμο στόχος. Δεν πάμε πετύχουμε κάτι τέτοιο σε 12-24 μήνες. Χρειάζεται όμως επαφές με τη Ρωσία. Δεν γίνεται αλλιώ. Η Ρωσία πρέπει να συμμετάσχει σε κάποιο συμπεφωνημένο αποτέλεσμα. Όποιο και θα είναι αυτό. Θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Εν τω μεταξύ, δεχόμενοι ότι η συλλογική ασφάλεια δεν προχωρά η Παναχωρή μάλιστα, τι κάνουμε. Είναι προφανές. Το ΝΑΤΟ είναι βασικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και του συστήματος Ευρωπαϊκής Ασφαλείας. Είναι το πλαίσιο εντός του οποίου συντονίζουμε τα στατιωτικά μας θέματα σε διεταντικό επίπεδο και θα χρειαστεί αυτό συνεχώς. Τίποτα δεν αποκλεί η αποτελεσματικότητα του ΝΑΤΟ να εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει αιτικές δυνατότητες και αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας όσον αφορά και τις επενδύσεις για την άμυνα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σεβαστά και να εφαρμοστούν. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα πρέπει τελικά να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Δεν αρκεί αυτό όμως. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι θεμελιώδης επαναξιολόγηση των σχέσεων των διατλαντικών Είπαμε, έχουμε υποχωρήσει όσον αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά στη διατλαντική κοινότητα, τα κράτη-μέλη δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, τα μέλη του ΝΑΤΟ και άλλε χώρε που θα ήθελαν να είναι εταίροι, μπορούμε να προχωρήσουμε. Να δημιουργήσουμε το είδο τη ασφαλεία και τάξη που θέλουμε και θέλαμε μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου. Και ελπίζουμε ότι σε κάποια φάση θα συμπράξουν και οι Ρώσοι συνάδελφοι. Οπότε, πού ερχόμαστε στο θέμα τη γειτονιά είναι σημαντικότατο να δούμε ποια είναι αυτή η πολιτική στις παρούσες περιστάσεις. Το είπαμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να λάβουμε υπόψη τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά στις σχέσεις με τη Ρωσία και τι μπορεί να κάνει η Ρωσία. Διότι έχει πολλά εργαλεία στη διάθεσή της, το απέδειξε. Μπορεί να δημιουργήσει και αντίθετα σενάρια, αντίπαλα σενάρια, επιπλοκές να εφαρμόσει ειδικέ πολιτικές. Οπότε η ανάπτυξη της πολιτικής γειτονίας αναπόφευκτα ε, συνδέεται με τη συζήτηση για τη σχέση με τη Ρωσία. Έτσι πρέπει να ειδωθεί. Δεν είναι ξεχωριστά θέματα. Τώρα να εστιαστούμε σε κάτι άλλο. Διαφοροποίηση μεταξύ προβλημάτων επιβολής του νόμου και ασφαλείας από τη μια και πολιτικών στρατιωτικών προβλημάτων απ' την άλλη. Αυτά είναι, ανήκουν στη σκληρή ασφάλεια, στο σκληρό πυρήνα της ασφάλειας. Μπορεί να παραθέσει κανείς σειράς παραδειγμάτων που δείχνουν ότι τα προβλήματα επιβολής του νόμου μπορούν να θεωρηθούν σαν προβλήματα στην αυτή η προσέγγιση φιλοσοφική δεν μπορεί να εφαρμοστεί και ίσως το κυβερνοχώρος είναι το πιο προφανές παράδειγμα. Αν δεν έχεις αποτελεσματικό σύστημα να εντοπίσεις την πηγή της επίθεσης δεν μπορείς να ξέρεις πια από πού προέρχεται η επίθεση και τι μορφή έχει η επίθεση του κυβερνοχώρου. Άρα για να βρούμε σωστή απάντηση στα προβλήματα ε, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και συνεργασία όσον αφορά τον κυβερνοχώρο. Μετά, υπάρχει και ατυχή στάση σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένοπλο έγκλημα που όλο και αυξάνεται. Τα εγκλήματα των συμμοριών, όπου τα άτομα ε, ε, εγκληματούν πιο εύκολα, έχουν πιο χαμηλό όριο και έχουν και όπλα που είναι και όλο και πιο θανατηφόρα. Όταν μιλάει κανείς με αστυνομικού, διαπιστώνει ότι σχετίζεται αυτό με την ησυχία τους για την ασφάλεια σε περιοχές όπως τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί έχουν μείνει πάρα πολλά όπλα και πυρομαχικά. Ανησυχούν επίσης για που μπορεί να αγοράσει κανείς από το διαδίκτυο διάφορα εργαλεία και τα ημιαυτόματα όπλα που είναι νόμιμα μπορεί να τα μετατρέψει με τα εργαλεία αυτά σε πλήρω αυτόματα που είναι παράνομα. Αυτά είναι θέματα που έχουν τεθεί επιτάπητος. Και αν δείτε τι γίνεται στα σύνορα, χωρίς να θέλει κανείς να κινδυνολογεί, βλέπουμε ότι έχουμε συγκρούσεις σε γειτονικέ χώρε Μήπως μπορούν να ξεχυλήσουν τα όπλα από εκεί, από την Ουκρανία Φερρυπίν, αλλού και από τη Μέση Ανατολή. Δεν πρέπει να είμαστε να κινδυνολογούμε, αλλά δεν μπορούμε να φυσικάζουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις μεταξύ τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας. Τι προσπαθούμε να πούμε στην έκθεση. Ότι τώρα ο άμεσος αντίκτυπος είναι σχετικά μικρός. Είχαμε τραγικά γεγονότα στο Παρίσι, στην Κοπενχάγη και αλλού, αλλά αν τα δει κανεί από ευρωπαϊκή σκοπιά είναι διαχειρίσιμα γεγονότα. Έχουμε και την εμπειρία του 2001. Συγκλονιστικό γεγονός μας έκανε να αντιδράσουμε με τρόπους ε, που τελικά απεδείχθησαν αντιπαραγωγικοί. Όταν βλέπουμε τώρα τις απειλές κατά της Ευρώπης πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη. Δεν μπορεί κανείς να φυσικάζει, το επαναλαμβάνω. Πρέπει να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Μην βρούμε απαντήσεις τώρα που εδράζονται επί άμεσης αντίδρασης εμφερμό που μπορεί να είναι κάτι αντιπαραγωγικό. Αυτό προσπαθούμε να πούμε. Στατιωτικές δαπάνες. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να τα εφαρμόσουν. Κάθε χρόνο δημοσιεύουν σχετικά στοιχεία. Υπάρχει συσχετισμός άμεσος μεταξύ αλλαγών στρατιωτικών δαπανών και εγκύτητα στη Ρωσία. Είναι σαφές. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έχει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα, επί παραδείγματι, αλλά η Ουκρανία αύξησε δραματικά τις αμυντικές δαπάνες για προφανέστατους λόγους. Αν δείτε λοιπόν το γενικό ανώτατο όριο των στατιωτικών δαπανών, των αμυντικών δαπανών, θα έλεγα ότι παραμένουν σταθερά αυτά όρια. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποίησεις περιφερειακές. Διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντιδρούν διαφορετικά ε, όσον αφορά τις απειλές που αντιλαμβάνονται. Ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Το πρόβλημα δεν είναι τα ποσά που δαπανώνται, αλλά ο τρόπος δαπάνης. Η Ρωσία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες κάθε χρόνο από το 99 και πιθανόν πριν από το 99, 15 χρόνια συνεχώς κάθε χρόνο σε πραγματικούς όρους αύξανε τις αμυντικές δαπάνες η Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια σημαντικότατες αυξήσεις όσον αφορά τα ποσοστά του ΑΕΠ της. Μετά από 15 χρόνια αυξήσεων, οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας αντιστοιχούν της Γαλλίας και της Γερμανίας αθρηστικά και προσπαθούν να διατηρήσουν και πυρηνικό δυναμικό, στατηγικά πυρηνικά όπλα, μη στατηγικά πυρηνικά όπλα, ε, προσπαθούν να προστατεύσουν τεράστια επικράτεια και έχουν και συμμετοχή σε πολλές επιχειρήσεις. Μάλλον εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις. Ξοδεύουμε πολλά χρήματα για την άμυνα. Δεν τα ξοδεύουμε σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άντωνη, αν δεν υπάρχουν σχόλια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της μελέτης. Να ευχαριστήσετε σας παρακαλώ και τους συναδέλφους σας, τους συναδέλφους από Λονδίνο και Παρίσι, από τα άλλα δύο Ινστιτούτα. Πολύ σημαντική βοήθεια για τον προβληματισμό μας και έξοχη εισαγωγή για την συνεδρίες επόμενης εβδομάδας στην Επιτροπή μας, όπου είπατε εκπρόσωπος η κυρία Μογκερίνη θα παρουσιάσει τις δικές της εκθέσεις που θα υποβάλει στο Συμβούλιο εν ώψη της αναθεωρήσεως της στρατηγικής της Ευρώπης για την ασφάλεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι το περιβάλλον άλλαξε πολύ από το 2003 μέχρι το 2008. Χρειάζονται νέες απαντήσεις, νέες κατευθύνσεις. Σε λιγότερο από 100 σελίδες μας δώσατε ε, κάποιες κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στο μέλλον τα προβλήματα και εδώ λίγη συνεδρίασή μας. Έχουμε συνεδρίσει σε το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με την αντιπροσωπεία μου. Εξέταση των σχέσεων με την Ουκρανία και εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Όσοι ενδιαφέρεστε είστε πρόσδεκτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη.